Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ε, ξεκινήσουμε. Θα εξετάσουμε την μύτη Έχουμε λοιπόν αυτές τις ε, ρυθμιστικές ε, προδιαγραφές ε, γιατί τώρα έχουμε εγκρίνει επιτέλους τις προδιαγραφές είμαστε όμως ακόμα στην φάση της εξέτασης και μπορεί ακόμα να υπάρξουν κάποιες αντιρρήσεις αλλά επειδή γνωρίζετε όλοι ακριβώς το πόσο μακροσκελής είναι αυτές οι διαδικασίες ε, συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, στην Κομισιόν, στο Κοινοβούλιο, εντός του Κοινοβουλίου. Την ε, συλλογική αυτή προσπάθεια για να βελτιώσουμε το κείμενο. Και επιφυλάσσουμε να μπούμε μετά σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι συνολικά το αποτέλεσμα αυτό είναι θετικό. Οπότε καμιά φορά χρειάζονται κάποιες περίπλοκες ε, κατασκευές, αλλά νομίζω ότι οι διάφορες ε, απαιτήσει και προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την Κομισιόν και να δώσω τον λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Μάρκος Φέμπερη. Προτιμάτε να ακούσετε, δεν ξέρω. Α, ωραία. Ξεκινάμε πρώτα με τον Μαρτέν Μερλέν. Καλώς ήρθατε και έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα το οποίο εξετάζεται σήμερα βεβαίως η πρόταση αυτή θέτει υψηλές προδιαγραφές για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και σημαίνει ότι θα υπάρχουν υψηλές απαιτήσει για την ταυτοποίηση των πελατών για να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη στο διαδικτυακό εμπόριο. Όμως το σημαντικότερο ζήτημα που τίθεται είναι η ασφαλής επικοινωνία μεταξύ τραπεζών και τρίτων μερών. Είχαμε εντατικές συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους, τα κράτη-μέλη και βεβαίως τους ευρωβουλευτές και θεωρούμε ότι θα βρεθεί έτσι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα όσα μας είπαν οι τράπεζες και οργανώσεις ε, καταναλωτών για το θέμα αυτό του καθαρίσματος των δεδομένων και βεβαίως των εταιριών FinTech που ανησυχούν ότι οι τράπεζες μπορεί να τους εμποδίσουν να προσφέρουν τις ε, καινοτόμες υπηρεσίες τους. Ακολουθήσαμε λοιπόν αυτό το οποίο μας είπε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ότι θα είναι υποχρεωτική η χρήση διεπαφών όταν ε, τις προσφέρουν οι τράπεζες. Αλλά υπάρχουν και διασφαλίσεις ε, για τις εταιρείες ε, FinTech και έτσι αν δεν πλήρούνται οι προδιαγραφές από το API e θα πρέπει να προσφέρουν μια εναλλακτική πλατφόρμα. Θεωρούμε λοιπόν τώρα άρα πως υπάρχουν πολύ ισχυρά κίνητρα έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά να αναπτύξουν κοινά API και να υπάρξει ένα νέο κύμα καινοτομία ε, οικονομικής ε, και χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας και έτσι θα μπορούν να οικοδομηθούν νέες ε, τέτοιες υπηρεσίες όπως ακριβώς συνέβη με τα έξυπνα τηλέφωνα. Οι πρώτες αντιδράσεις των εταιριών ήταν πολύ θετικές και των εταιριών FinTech και των τραπεζών και τώρα θέλουν να αρχίσουν να συνεργάζονται σε πρότυπα διαπαφής ε, και η Κομισιόν με την Κεντρική Τράπεζα δημιουργούν μια ομάδα που θα διευκολύνει ακριβώς ε, την επαφή μεταξύ των δύο αυτών ε, μέρων. Η πρώτη συνεδρία θα γίνει την Δευτέρα. Οι συμμετέχοντες στην αγορά μας λένε ότι χρειάζεται βεβαιότητα νομική το συντομότερο δυνατόν, οπότε ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να δημοσιευτεί αυτή η απόφαση στην ε, επίσημη εφημερίδα, ελπίζουμε τον Μάρτιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, Dirk Aubrich. Ε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στο ένα λεπτό που μας έχετε δώσει. Ευχαριστώ και την ε, Κομισιόν για την πρόοδο που έκανε στο θέμα. Εμείς δεν είμαστε τόσο πεπισμένοι όσο η Κομισιόν για λόγους ουσιαστικούς και διαδικαστικούς. Η διαδικαστική είναι το ότι η Κομισιόν απέρριψε κάποιες από τις ανησυχίες ή δεν τις δέχτηκε ανησυχίες που είχαμε εκφράσει στην γνωμοδότησή μας τον Ιούνιο, που είναι βεβαίως δικαίωμά της, αλλά όταν εγκρίναμε την πρόταση τον Νοέμβριο είδαμε ότι υπήρχαν κάποιες επιπλέον απαιτήσει τι οποίες δεν γνωρίζαμε και θα θέλαμε να έχουμε την δυνατότητα να τις ε, σχολιάσουμε όπως απαιτεί ο κανονισμό μας. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ε, ένα προηγούμενο που δεν είχαμε δει στα άλλα 148, σε άλλες 148 τεχνικές προδιαγραφές. Μία ανησυχία θα αναφέρω μόνο, η οποία αφορά τον βαθμό στον οποίο ε, η Κομισιόν μίλησε για μια ισορροπημένη λύση και το πώς ε, το screen scraping θα πρέπει να επιτραπεί και από τις δύο πλευρές. Εμείς έχουμε ελαφρώς διαφορετική άποψη μετά από τις επαφές μας με τον κλάδο, αλλά αν ισχύει όντως ότι η εντύπωση της Κομισιόν ε, του, ή του Κοινοβουλίου είναι ότι έχουμε μια ισορροπημένη άποψη, είναι, αυτό οφείλεται στο ότι η τεχνική προδιαγραφή δεν έχει καθορίσει το εάν θα επιτρέπεται ή όχι το screen scraping. Είναι μια πολιτική απόφαση η οποία παραπέμπεται ε, στο μέλλον. Γιατί η τεχνική προδιαγραφή λέει ότι αυτό θα το αξιολογήσει η αρμόδια αρχή με βάση την αξιολόγηση της διαπαφής. Κάτι το οποίο δεν είναι πρόβλημα να το κάνουν οι αρμόδιες αρχές γιατί βεβαίως είναι επόπτες αλλά θα πρέπει να κρίνουν το εάν είναι και αξιόπιστες ε, οι ίδιοι αυτές. Αυτό όμως είναι μια αξιολόγηση πληροφορικής για το οποίο δεν έχουν τα προσόντα και την αρμοδιότητα να το κάνουν. οι εθνικές εποπτικές αρχές και επίσης θα πρέπει να κρίνουν τις υποδομές ε, της ε, κάθε συγκεκριμένης τράπεζας. Οπότε μιλάμε για χιλιάδες τέτοιες αξιολογήσεις. Υπάρχουν 6.000 τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλήγοντα λοιπόν, στην αξιολόγηση αυτή πρέπει να πληρούνται κάποιοι όροι σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή και κάποια από αυτά μας ανησυχούν εμάς και τις εθνικές αρχές γιατί υπάρχει τώρα το βάρος της συμμόρφωσης ε, και ένας από τους όρους λέει ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη το εάν ε, οι διαπαφές που παρέχονται από την τράπεζα ικανοποιούν ε, TPP, ε, δηλαδή η απόφαση αυτή εξαρτάται από το εάν ε, κάποιοι άλλοι η ε, TPP είναι ικανοποιημένοι από αυτήν την διαπαφή το οποίο είναι ασυνήθιστο νομικά και νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Έχουμε νομίζω ένα-δύο μήνες να το σκεφτούμε, αλλά θα έχουμε δύσκολες συζητήσεις σε 6 ή 18 μήνες για κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποια σχόλια, αλλά καταρχήν θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για αυτά τα οποία είπε. Έχουμε έντονες συζητήσεις που γίνονται όχι μόνο εδώ αλλά και διμερός και νομίζω ότι καταφέραμε να βρούμε έναν καλό συμβασμό που θα επιτύχει τους στόχους του PSD2, δηλαδή το άνοιγμα των σχετικών αγορών πληρωμών με υψηλή προστασία των καταναλωτών. Και τα μηνύματα που λαμβάνω εγώ από τους συμμετέχοντες στις αγορές είναι ότι πρόκειται για έναν ισορροπημένο συμβιβασμό. Γι' αυτό είμαι και ικανοποιημένος, όπως ε, και η Κομισιόν άλλωστε. Έχω δύο ερωτήσεις. Ε, η τεχνική προδιαγραφή προβλέπει ότι οι εθνικές αρχές ε, μπορούν να δώσουν απαλλαγή από την υποχρέωση να υπάρξει ένας μηχανισμός backup αρκεί να πληρούνται κάποια κριτήρια και τα κριτήρια είναι ότι θα πρέπει να έχει περάσει ο μηχανισμός μια δοκιμή τριών μηνών σε πραγματικές συνθήκες και να είναι οι χρήστες ε, ικανοποιημένοι. Αλλά τι θα γίνει αν η τράπεζα ή κάποιος τρίτος ε, δεν είναι ικανοποιημένος ή εάν οι δύο αξιολογήσεις αποκλίνουν. Υπάρχουν κάποια κριτήρια με τα οποία μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα οδηγηθούμε σε κάποιο είδους αρμπιτράζ και τέλο ε, όσον αφορά τα stress test προβλέπεται ότι οι εθνικές αρχές θα έχουν την εποπτεία και μάλιστα με μια συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία θα αναλάβει την αξιολόγηση αυτή. Πώς το φαντάζεστε ένα τέτοιο stress test, κάθε πότε θα γίνεται, ποιες λειτουργίες ε, θα εξετάζονται, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές ή τεχνικές προδιαγραφές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για να διασφαλίσουμε ότι τα stress test των εθνικών αρχών θα είναι συγκρίσιμα. Όχι η μία αρχή να κάνει στην χώρα Α ε, την ε, εξέταση αυτή με διαφορετικά κριτήρια από τη χώρα Β. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λουδβίξον. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε πως η πρόταση αυτή της Κομισιόν για τα τεχνικά πρότυπα για τις ασφαλείς επικοινωνίες είναι μια εξαιρετική ε, ένα εξαιρετικό συμβιβασμό μεταξύ των συμφερόντων των εταιριών FinTech και των παραδοσιακών τραπεζών. Θα είναι υποχρεωτικά όλα αυτά όταν τη στιγμή τη ταυτοποίηση από τι τράπεζε, αλλά για να το πετύχουμε θα πρέπει η τεχνολογία να είναι στη θέση τη και σωστή. Και το καλό θα είναι οι TTP να μπορούν να κάνουν κάποιε πληρωμέ, ακόμα και αν η διεπαφή αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα. Τώρα, στις προτάσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σας πω πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει πολλά για να έχουμε ισότιμους κανόνες αγοράς στο θέμα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και με τον τρόπο αυτό θα έχουν ε, πρόσβαση στις πληροφορίες λογαριασμού των πελατών ή TPP μόνο στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Και γι' αυτό είμαι υπέρ ε, των τεχνικών προδιαγραφών RTS με τον τρόπο που έχουν αυτές διατυπωθεί. Thank you. Um, other colleagues. Άλλοι συνάδελφοι. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Να γνωρίζω πως από τη δική μου οπτική γωνία. Η λύση αυτή δεν είναι τέλεια και πρέπει να σας πω πως με τις προτάσεις που είχε κάνει η EBA εγώ τουλάχιστον ήμουν σύμφωνος ε, βέβαια αυτό δεν εκπροσωπεί όλο το κοινοβούλιο και τώρα έχουμε και τις εξαιρέσεις ε, που μας οδηγούν στο fallback, ε, τις τεχνικές δυνατότητες που οδήγησαν στο συμβιβασμό, ε, τις διαπαφές κτλ. Εν πάση περιπτώσει αυτά θα πρέπει να τα σεβαστούμε και σε σχέση με το προηγούμενο κείμενο το οποίο είχε παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώ ότι η εξαίρεση που δίνεται εδώ είναι μια βελτιωμένη μορφή της πρότασης. Βεβαίως προκύπτουν μια σειρά θέματα για το πώς ακριβώς θα λειτουργεί Προφανώς υπάρχει ένας ρόλος κομβικός τον οποίο αναλαμβάνει η EBA έτσι ώστε να εξασφαλίσει πως οι εθνικές αρχές ε, κάνουν μια παρόμοια ερμηνεία τη στιγμή που ε, αξιολογούν την ποιότητα ε, της διαπαφής για να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα εξαίρεσης γιατί οποιαδήποτε διαφορά στην ερμηνεία μπορεί να οδηγήσει σε κακή λειτουργία της ε, ε, εσωτερικής αγοράς στη στιγμή αυτών των πληρωμών και επίσης οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν την επαλήθευση ε, για παράδειγμα των πρωτοκόλων για τις πληρωμές που έχουν εξαιρεθεί και τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 17 και άλλα τέτοια καθήκοντα, τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τεχνικών προδιαγραφών για τις διαπαφές άρθρο 30 σημείο 6 της παρακολούθησης των τεχσταντοχής μέσω των διαπαφών το 32 δύο, οπότε είναι πολλά. Και για να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο εποπτικής σύγκλησης και να εξασφαλίσουμε πως έχουμε προστασία του καταναλωτή, είναι σημαντικό να έχουμε την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ αρμοδίων αρχών, της EBA, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εμπλεκομένων. Και τέτοιου είδους εποπτική σύγκληση προβλέπεται έτσι ώστε να κάνουμε μία ε, ένα streamlining αυτών των τεχνικών προδιαγραφών RTS για παράδειγμα, ε, για την επαλήθευση της συγκεκριμένη ε, διεπαφής και τη διασφάλιση της ασφάλειας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής. Για όλα αυτά, λοιπόν, Γιατί βέβαια δεν θα πρέπει να είναι ο ανταγωνισμό τον οποίο θα πρέπει να ικανοποιήσουμε, ε, ο ανταγωνιστή τον οποίο θα πρέπει να ικανοποιήσουμε. Θα πρέπει οι αρμόδιε αρχέ, έτσι το διαβάζω, θα βοηθήσουν αυτού οι οποίοι δείχνουν μια ε, ισορροπημένη ε, προσέγγιση και δεν αφήνουν τους λόγους του ανταγωνισμού να πριτανεύσουν έτσι ώστε η διαδικασία αυτή να γίνει μια ζούγκλα Χρειαζόμαστε ισορροπημένη, ε, στέρεη διαδικασία με καλή σύγκληση. Βέβαια χρειάζονται πόροι και κατανοώ τη δυσκολία εδώ, αλλά αυτό είναι μια προϋπόθεση, εάν επιθυμούμε, αυτές οι δύο επαφές να, να αποτελέσουν το πρότυπο που θα είναι καλές, ανοιχτές, προσβάσιμες από όλους, αλλά παράλληλα ασφαλείς και προσφέρουν το επίπεδο εκείνο ασφάλειας το οποίο επιθυμούμε. Οπότε η εξαίρεση θα πρέπει να δίδεται με έναν ε, τρόπο που θα ε, αποδεικνύει πως υπάρχει συνοχή και ε, δικαιοσύνη και θεμητός ανταγωνισμός και όχι για να εξασφαλίσουμε τη θέση του χ ή του ψ ανταγωνιστή στην αγορά. Και το λέω γιατί για να, για να λειτουργήσει αυτός ο συμβιβασμός πολλά μένουν να γίνουν και πολλά πρέπει να εφαρμοστούν και γι' αυτό στρέφομαι προς την EBA και την Κομισιόν να μου πούν τα θέματα αυτά πώς θα τα αντιμετωπίσετε, πώς θα εξασφαλίσετε, πώς θα πετύχετε αυτό το στόχο. Thank you. Thank you, Chairman, for this. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια αυτά κύριε Πρόεδρε και θα δώσω μία σύντομη απάντηση. Όπως είπα και στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις εμείς αυτό που κάναμε ήταν να δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών και των εταιριών FinTech που θα ξεκινήσει από Δευτέρα να δουλεύει και πιστεύουμε πως εδώ θα εκεί μάλλον θα αποφασιστούν οι ε, πρακτικές λεπτομέρειες και θα οριστούν εκεί έτσι ώστε αυτά τα, αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές και τα RTS να εφαρμοστούν με τον κατάλληλο τρόπο. Θα τους δοθούν έξι μήνες και βεβαίως θα στηριχθούν από την Κομισιόν και από την ΕΚΤ και ελπίζουμε πως και η EBA θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν επιπλέον κάνει τη δουλειά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρόλα αυτά χρειάζονται και άλλες τεχνικές προδιαγραφές, για να πετύχουμε τα θέματα των τεχνικών, να πετύχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε στις τεχνικές προδιαγραφές. Ναι. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ερωτηματολόγιο, ένα Q&A της CBA προς υποστήριξη. Τώρα, για το ποιος πρέπει να αξιολογήσει την ποιότητα των διεπαφών, Πιστεύουμε πως αυτός είναι ο ρόλος των εθνικών αρχών ε, υπό την αιγίδα της EBA με τρόπους στην πράξη που ακόμα μένουν να αποσαφινιστούν και για το κατά πόσο αυτά τα stress tests ε, μας αφορούν πιστεύω πως θα πρέπει οι παίκτες στην αγορά να είναι σε θέση να συμφωνήσουν πώς αυτά τα τεστ αντοχής θα λειτουργήσουν, θα περιγραφούν και εκεί πάλι αν κριθεί απαραίτητο και μετά αυτή την πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ εταιριών FinTech και ε, τραπεζών τότε θα μπορούσε να παρέμβει η EBA και να περιγράψει πώς αυτά τα τεστ αντοχής θα λάβουν χώρα. Σε δέκα δευτερόλεπτα να σας πω πως η Κομισιόν είπε πολλά τα οποία και εμείς θα στηρίξουμε. Το κομβικό ζήτημα είναι το να κλείσουν τεχνικές λεπτομέρειες γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρχει εταιρική σαφήνεια στο θέμα των τεχνικών προδιαγραφών, τα θέματα που θα προκύψουν και θα πρέπει η EBA να αντιμετωπίσει μέσα σε 6, 12, 18 μήνες θα είναι ατελείωτα και δεν έχουμε τους πόρους. Μάρκου, μία σύντομη παρατήρηση. Χαίρομαι για την πρόοδο που έχει σημειωθεί και κατανοώ και ποιο είναι το πλαίσιο με στο οποίο ε, εργαζόμαστε. Βλέπω ότι εδώ χρειάζεται και η συμμετοχή της ΕΚΤ και η συνεργασία αυτή νομίζω ότι πραγματικά ανταποκρίνεται σαν όσα έχουμε στην καρδιά της νομοθεσίας μας, η οποία δεν είχε σκοπό να προστατεύσει τις τράπεζες ούτε τις fintech. Είχε σκοπό να προστατεύσει τον καταναλωτή. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως μπορεί να συγκεράσει τις δύο πλευρές ε, προς όφελος του καταναλωτή. Γι' αυτό τα έχουμε όλα αυτά. Και νομίζω πως ο συμβιβασμός που πετύχαμε είναι καλός και ισορροπημένος. Πολύ ωραία. Νομίζω πως ε, είναι τεράστιο το καθήκον για τις ε, αρμόδιες εθνικές αρχές και για την EBA και θα πρέπει αυτά να τα λάβουμε υπόψη όταν θα γίνει ο συνηθισμένος διάλογος για το θέμα των πόρων. γιατί πρέπει να μπορέσουμε εμείς να παραδώσουμε και εσείς επίσης αυτά τα οποία μας ζητάνε. Θέλουμε αυτά τα, αυτές οι διαπαφές να αποτελέσουν το πρότυπο. Δεν θέλουμε το fallback. Η καλύτερη λύση είναι οι διαπαφές που λειτουργούν. Αλλά αυτό χρειάζεται ελέγχους, επαλήθευση. Να μην έχουμε κατάχρηση αυτών να μην ε, κάνουν οποιαδήποτε κατάχρηση και τα δύο μέρη, δηλαδή και αυτοί που χρησιμοποιούν την υπηρεσία, οι πελάτες δηλαδή, και αυτοί που την προσφέρουν. Και να μην μποϊκοτάρουν, για παράδειγμα, κάποιοι οποίοι θέλουν το screen scraping ως προτιμούμενη λύση. Ε, ε, Αυτά. Και η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο. Κατανοώ βέβαια το τεράστιο βάρος για την EBA και για τις εθνικές αρχές. Όπως είπα, προ... τιμούσα το αρχικό RTS, τεχνικές προδιαγραφές που είχατε παρουσιάσει, αλλά εδώ που φτάσαμε είναι και μια ευκαιρία. Να έχουμε μια εποπτική αρμοδιότητα η οποία θα είναι ισορροπημένη και που θα δίνει τα, παρά, τα απαραίτητα εχέγγυα έτσι ώστε να μην ασχολούνται μόνο με το θέμα αυτό οι εμπλεκόμενοι αλλά να εξασφαλίσουμε πως όλοι θα ακουστούν και πως όλα θα γίνουν με δίκιο τρόπο. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία, θα σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε και χαίρομαι που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως αν είναι απαραίτητες οι κατευθυντήριες γραμμές, αν χρειάζεται Q&A, τότε θα επιστρέψουμε και αν κάτι δεν λειτουργήσει θα το φτιάξουμε. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία και για να δούμε αν χρειάζονται κάπου διορθώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο θέμα που αφήνω σε σένα Μάρκους. Uh, Μάλιστα. Το επόμενο θέμα το θέμα της ε, σε MIFID με τις, για τις τρίτες χώρες. Ποιος είναι εδώ από την Επιτροπή Δεν ξέρω ποιος είναι εδώ από την Επιτροπή, δεν έχω δει κανέναν. Α, τώρα σας είδα, ναι, συγγνώμη. Τώρα βλέπω την ε, ομάδα MIFID. ευχαριστώ που ήρθατε. Έχετε το λόγο. Thank um, Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσουμε για τις ε, αποφάσεις αντιστοίχησης που λάβαμε καθώς και για την ευκαιρία να μπορέσουμε να σας κάνουμε μια σύντομη ενημέρωση για το τι έχει συμβεί μετά από τις αποφάσεις αντιστοίχησης που ελήφθησαν. Ήδη αυτές οι αποφάσεις ισχύουν εδώ και ε, τρεις εβδομάδες και συζητήσαμε με τους ρυθμιστές της χώρας όπου ε, ε, ισχύει η αντιστοιχεία για να ελέγξουμε τι ε, συνέβη στην πράξη εφόσον εκδόθηκαν αυτές οι αποφάσεις και έχουμε και κάποια αρχικά πορίσματα να μοιραστούμε μαζί σας. Για να ανακεφαλαιάσω, ε, μιλήσαμε για τα παράγω... την εμπορία παραγόγων και μετοχών. Στα παράγωγα πρόκειται για ένα πρόγραμμα αμοιβαίας αναγνώρισης, δηλαδή χορηγούμε αντιστοιχεία για τη συμμόρφωση προς την εφαρμογή ε, της, ανταλλαγή και του και των υποχρεώσεων ε, ε, εμπορίας και τούμπαλιν. Έτσι έχουμε λοιπόν μία δικαιοδοσία αυτή τη στιγμή που αναγνωρίζεται, είναι η ΕΠΑ, διότι βεβαίως η ΕΠΑ όπως γνωρίζετε έχει υποχρέωση εμπορίας για ορισμένα παράγωγα από το 2013 έχουμε αναγνωρίσει και μία ολόκληρη σειρά βάσεων εκτέλεση ΣΟΠΑ στη ΣΥΠΑ ε, έχει αναγνωριστεί και η δική μας ε, αντίστοιχη αγορά χρεογράφων και το Αμερικανικό STC έχει εκδώσει μία ε, διαταγή εξαίρεσης ώστε οι Αμερικανοί μπορούν να ε, χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκά ε, χρηματιστήρια για τις δικές τους συναλλαγές. Πρόκειται για εξαιρετικά ρευστά μέσα. Οι πρώτες ε, εμπειρίε είναι αρκετά εθαρρυντικές, το σύστημα λειτουργεί. Έχουμε μόνο κάποια αναπομείναντα θέματα που πρέπει να τα ρυθμίσουμε και αυτά κυρίως οφείλονται στο γεγονός ότι έχουμε το πιο, πιο καινούριο σύστημα από τις είπα. Όταν έγινε λοιπόν η αντιστοιχεία, η ΕΠΑ ήδη είχε, είχαν μια λίστα 12 ε, καταστάσεων ε, δυνατότητας ε, swap ενώ οι δικές μας λίστες έμπαιναν σταδιακά online. Έχουμε έναν αρχικό κατάλογο με ευρωπαϊκά φόρα αλλά θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά καθώς μπαίνουν online και νέες δυνατότητες ευρωπαϊκές. οι, όσοι χρησιμοποιούν τώρα τις ευρωπαϊκές ε, πλατφόρμες χρησιμοποιούν, ε, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις αμερικανικές δυνατότητες διάδοσης και εμείς ε, πρέπει να, να, ενεργήσουμε έτσι ώστε να αναγνωρίζεται και το δικό μας σύστημα αναφορών το οποίο ωστόσο πράγματι είναι κάπως διαφορετικό. αλλά δεν αμφισβητεί την αμοιβαία αναγνώριση την ίδια. Έπειτα έχουμε κάποιες αναπομείνασες ε, δικαιοδοσίες ε, στο μέτωπο των ε, παραγόγων όπου δεν υπάρχει πλήρης αναγνώριση Σιγκαπούρη και Αυστραλία. Μόλις θα θεσπιστούν τέτοιες εμπορικές υποχρεώσεις και χρεόγραφα θα αναγνωριστούν και τα ευρωπαϊκά, οι ευρωπαϊκές δυνατότητες για την εκτέλεση αυτών. Τώρα, για τις μετοχές, έχουμε αναγνωρίσει όσον αφορά την υποχρέωση εμπορία μετοχών την ΣΥΠΑ, την Ελβετία, το Χονγκ και την Αυστραλία και υπάρχει μια επιπλέον απόφαση που προετοιμάζεται και αφορά την Νότιο Αφρική. Και ελπίζουμε πως θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία στο εγγύς μέλλον. Με αυτές τις δικαιοδοσίες λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι καλύπτουμε όλες τις δικαιοδοσίες που έχουν ε, εκδόσεις μετοχών που ε, ε, εμπορευόμαστε και ανταλλάσσουμε και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Εάν δηλαδή η έκδοση συγκεκριμένης δικαιοδοσίας χρησιμοποιείται στην Ένωση, ε, ή όχι. Έχουμε καλύψει λοιπόν το διπλό σενάριο, τις διπλές διπλά εντεταγμένες εταιρείε ε, με τις ίπα το Χονγκ Κόνγκ και την Αυστραλία και τώρα έχουμε να κάνουμε και με τη δίκτυα SMI της Ελβετίας, ε, ο οποίος χρησιμοποιείται πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η απόφαση ήταν πολύ σημαντική και απαραίτητη. Έχουμε ακόμα μετοχές που είναι διπλά καταχωρημένε ε, καταχωρημένες και στην Ένωση και στις ΕΠΑ και πρέπει να εγκριθεί και αυτό το πακέτο. Έχουμε και ένα μικρό αριθμό, δύο-τρεις ε, διπλές καταχωρήσεις με το Χονγκ Κόνγκ και με την Αυστραλία. Ωστόσο, για να είμαστε απόλυτα βέβαιοι, αναγνωρίσαμε και αυτές τις δυο δικαιοδοσίες. Πρώτα αποτελέσματα λοιπόν, τι έγινε μετά από τις αποφάσεις αντιστοιχίας, άλλαξε κάτι όσον αφορά τα, τα, ε, τις μορφές εμπορίου. Θα ξεκινήσω με την Ελβετία, η οποία έχει μεγάλο ογκό, κατέχει μεγάλο ογκό εδώ στην Ένωση, αλλά και στο δικό της χρηματιστήριο αρχικά είμαστε 50-50, κάποιες περιπτώσεις είναι 70-30 και ή 40-60 και αρχικές συνέπειες αυτής της απόφασης αντιστοιχής ήταν ότι λόγω των μεγεθών έχει υπάρξει μετακίνηση προς τις ελβετικές πλατφόρμες. Το χρηματιστήριο ΣΥΚΣ λοιπόν μεταφέρθηκε από το 61% μάλλον αυξήθηκε στο 71% μετά την αντιστοίχηση. Και οι ευρωπαϊκές πλατφόρμες οι οποίες είναι καταχωρημένες που είναι συνιστώσεις του SMI 20 χάσανε λίγο 2 με 3% σε κάθε ε, χρηματιστήριο. Επειδή όμως τα μεγέθη στην Ελβετία είναι πιο στενά και με μεγαλύτερος όγκος, συνεχίζεται ε, κάποια ροή όγκου προς τις ελβετικές ε, ε, τα ελβετικά χρηματιστήρια. Χρειάζεται βέβαια να προσαρμοστούν οι δείκτες, οι ευρωπαϊκοί, με τους ελβετικούς, ώστε να υπάρχει ισότιμο πεδίο. Τέλος, σε ένα άλλη δικαιοδοσία που έχουμε κάποια πρωταπορίσματα, πορίσματα, είπα, όπου έχουμε κάπου 12 εταιρείες που είναι καταχωρημένες και στις ΕΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις ΕΠΑ είναι δευτερογενής ε, καταχώρηση και το εμπόριο σε θέματα όγκου είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι αυτό που γίνεται στην Ευρώπη. Το πρώτο μας πόρισμα είναι ότι στις ΕΠΑ δεν υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στις ε, ροές Καταρχάς δεν έχουμε αύξηση στις ροές στις συγκεκριμένες μετοχές. Για να, να είμαι πιο ακριβής, έχουμε 14 στην υποχρέωση ε, Ένωσης και 4 στην Αμερική. Και βλέπουμε ότι οι συναλλαγές σε αυτές τις μετοχές μειώθηκαν μετά από την αντιστοίχηση. Δεν θα πει αυτό ότι αυτό οφείλεται στη ΜΥΦΙΔ. Ο συνολικός όγκος των, μετοχών, των συναλλαγών μάλλον σε μετοχές στη ΣΥΠΑ μειώθηκε στις τρεις πρώτες εβδομάδες του 2018 σε σχέση με τις τρεις πρώτες εβδομάδες του 17. Ένδο και έξω χρηματιστηριακές συναλλαγές παρέμειναν σταθερές ε, ωστόσο στη ΣΥΠΑ, οπότε και μετά την αντιστοίχηση δεν υπήρξε μεγάλη μετακίνηση στις συναλλαγές για τις ε, μετοχές οι οποίες είναι καταχωρημένες και στην Ένωση και στις ΗΠΑ. Εν γέννη λοιπόν πιστεύω ότι καλυπτόμεθα με τους πιο σημαντικούς μας ε, εταίρους Δηλαδή όλες οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλο όγκο συναλλαγών ε, στην Ένωση καλύπτονται από τις αντιστοιχήσεις. Ε, όπως σας είπα, προς την Ελβετία έγινε μετακίνηση και σας εξήγησα για ποιους λόγους. Αλλά στις ε, ΗΠΑ, όπου δεν έχουμε πολύ μεγάλη επικάλυψη, δεν υπήρξαν αλλαγές. γιατί Παραμένουν σταθερά τα πράγματα στο 66% στο χρηματιστήριο και 44% εκτός χρηματιστηρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωστερμαν από την ΕΣΜΑ και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που εξετάζετε τις αποφάσεις αυτές του Μηφιντ μα δεν έχει κάποιον επίσημο ρόλο στην διαδικασία ισοδυναμίας αλλά ευχαριστώ να σας πούμε τις απόψεις μας για τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί συγκεκριμένα θα αναφερθώ στην υποχρέωση εμπορίας μετοχών και μετά βέβαια θα περάσω και στις ε, τρίτες ε, χώρες ε, και στα παράγωγα και στο πλαίσιο ισοδυναμίας. Ξεκινώντας με τις μετοχές μπορώ να επιβεβαιώσω πως πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει και ανησυχεί τις χώρες εκτός της Ένωσης. Γεγονός είναι πως περισσότερες μετοχές που έχουν την κύρια πηγή ρευστότητα σε τρίτες χώρες ε, είναι αντικείμενα εμπορία και εντός της Ένωσης και εμπίπτουν στην MIFID 2. Υπήρχε λοιπόν βάσιμες ανησυχίες από ρυθμιστικές αρχές τρίτων χωρών όταν τους επηρέαζε η MIFID 2 και πιθανώς υπήρχε κίνδυνο αποκοπή ε, των Ευρωπαίων επενδυτών κατά το οποίο θα επηρέαζε την ρευστότητά του και βέβαια θα υπήρχαν και πιθανά ε, πιθανές συνέπειες ε, γι' αυτό χαιρόμαστε για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε αποφάσεις ισοδυναμίας για διάφορες δικαιοδοσίες όπως εξηγήθηκε ήδη και έτσι συνεχίζεται η πρόσβαση των Ευρωπαίων επενδυτών στις παγκόσμιες αγορές. Για να εξηγήσουμε λοιπόν την παγκόσμια ισχύ της MIFID 2 θα ήθελα να σας πω μια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η ΕΣΜΑ εκτός αυτού του πλαισίου. Πρόκειται για την υποχρέωση για όλα τα μέσα τα οποία είναι αντικείμενα εμπορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για όσα έχουν απλά οριακές συναλλαγές εντός της Ένωσης. Αυτό σημαίνει πως οτιδήποτε γίνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια επενδυτική εταιρεία θα πρέπει να υφίσταται έλεγχο ως μια συναλλαγή OTC, όμως αυτό θα ήταν υπερβολικό βάρος για τις εταιρείες αυτές οι οποίες έχουν έδρα σε τρίτες χώρες. Γι' αυτό Κοιτάμε ακριβώς ως έσμα το εάν υπάρχει επαρκής διαφάνεια στην τρίτη χώρα, οπότε να μην χρειάζεται να ξαναγίνει το ίδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία μας αυτή επίσης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και έχουμε ε, ακούσει τις αντιδράσεις από 100 περίπου ε, δικαιοδοσίες. Τώρα θα περάσω στα παράγωγα, όπου πρώτα απ' όλα είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι εγκρίθηκε εγκαίρως η σχετική τεχνική προδιαγραφή και έχει αρχίσει να ισχύει από 18 Ιανουαρίου και βεβαίως ε, είναι σημαντικό η εφαρμογή να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην διεθνή διάσταση εμείς ε, ακριβώς έχουμε δώσει αυτή την διεθνή διάσταση στην τεχνική προδιαγραφή και έχουμε εξετάσει τις υποχρεώσεις που υπάρχουν σε άλλες χώρες, ειδικά στη ΣΥΠΑ. Γι' αυτό Επίση, καλωσορίζουμε το ότι ενέκρινε η Κομισιόν μια απόφαση ισοδυναμία με τις ΕΠΑ στο πλαίσιο της ε, υποχρέωσης αυτής εμπορίας παραγόγων κάτι το οποίο θα επηρεάζει σαφώ λιγότερες χώρες από ότι η σχετική υποχρέωση για τις μετοχές ε, θα πρέπει να δούμε και τις μεγάλες δικαιοδοσίες σε αυτό το θέμα. Κλείνοντας ε, θα κάνω μια γρήγορη ανασκόπηση του γενικότερου καθεστώτος ισοδυναμίας στη MIFID 2 προφανώς έχει μεγάλη σημασία και στο πλαίσιο του Brexit η επαφή με τρίτες χώρες ίσως γίνει ακόμη πιο σημαντικό το θέμα στο μέλλον. Το καθεστώς ισοδυναμίας της MIFID 2 είναι πολύ πολύπλοκο και αποσπασματικό Γι' αυτό θεωρούμε ότι εάν παρουσιαστεί ευκαιρία το καθεστώς αυτό ίσως αξίζει να επανεξεταστεί και είμαστε στην διάθεσή σας για τυχόν σύμβουλες. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στην διαπραγματευτική ομάδα που θα το, το δώσουμε τώρα στον εισηγητή που θα μιλήσει τη μητρική του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την γενική εικόνα που μας δώσατε. Έχουμε την συμφωνία αυτή ισοδυναμίας με τις ε, ΗΠΑ, Αυστραλία και Ελβετία. Ακριβώ ε, απολογισμός είναι κάπως ε, παίρνει χρόνο βεβαίως τι αποτελέσματα είχε στα παράγωγα αν μπορεί επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει τα καθήκοντά της με έναν κατάλογο δικαιοδοσιών και με ποιες ακριβώς δικαιοδοσίες έχουμε την ε, αναγνώριση αυτή και αν θα περιμένουμε και περαιτέρω τέτοιες ε, συμφωνίες. Ελπίζω να μην είναι τους σοσιαλιστές εκεί που μιλάνε. Θα ήθελα επίσης να μάθω ποιες ε, εμπειρίες είχε η Κομισιόν όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για νέες συμφωνίες ισοδυναμίας και επίσης αν έχει τους απαραίτητους πόρους για να κρίνει κάτι τέτοιο και το ρωτώ αυτό λόγω της συμφωνίας με τις είπα και συγκεκριμένα για το θέμα ε, ποιο είναι το αστείο πείτε μας και εμάς να γελάσουμε η κατάταξη των λεγόμενων εναλλακτικών συστημάτων ε, τεχνικών προδιαγραφών γιατί είχα την εντύπωση πως ένα μεγάλο κομμάτι των, των ισοδυναμιών αυτών τελικά θα ήταν αυτές τις οποίες είχε αποφασίσει η Επιτροπή Κεφαλαίου αγορά των ΙΠΑ, τις οποίες απλώς αντέγραψε η Κομισιόν. Και βεβαίως λογικό θα είναι να περιμένουμε να μην ε, περιέχουν οι δηλώσεις τρίτων χωρών λανθασμένες ε, πληροφορίες. Επίσης, ε, από πλευράς Κομισιόν, ο κύριος Μαγιόρ είχε απευθύνει μια επιστολή τον Νοέμβριο που αφορούσε κάποια προβληματικά σημεία του καθεστώτος ισοδυναμίας ε, τρίτων χωρών, ότι δηλαδή δεν υπάρχει ένα επανευρωπαϊκό τέτοιο καθεστώς για πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, δεν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει μία βραχυπρόθεσμη πάυση της ε, εμπορίας ε, παραγόγων και βεβαίω υπάρχουν και όλα εκείνα τα καθεστώτα τρίτων χωρών τα οποία έχουν μια πιο, ε, ένα πιο ελαφρύ ρυθμιστικό καθεστώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και η Κομισιόν πώς εκτιμά την κατάσταση και με συγχωρείτε που αναφέρω ξανά το θέμα. Υπάρχουμε μια χώρα που είναι αυτή τη στιγμή εντός της Ένωσης αλλά προσεχώς θα γίνει τρίτη χώρα και όταν διαπραγματευτήκαμε το MIFID 2 κανείς ε, δεν είχε την ε, δυνατότητα να σκεφτεί ότι θα φύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το καθεστώς ε, τρίτων χωρών δεν δημιουργήθηκε ότι η μεγαλύτερη έχοντας κατά νου ότι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χρηματαγορά θα γίνει ξαφνικά τρίτη χώρα. Οπότε θα ήθελα να μάθω πώς ε, βλέπουν η Κομισιόν και η ΕΣΜΑ τις μελλοντικές σχέσεις με τα καθεστώτα τρίτων χωρών και αν απαιτείται εδώ πέρα κάποια αλλαγή. Ειδικά δεδομένων των όσων αναφέρει η Μήφυρ στα άρθρα 35 και 36. Να συνεχίσω η Περμάς θέλει να μιλήσει για τους σοσιαλδημοκράτες. Νομίζω πως τα βασικά τα είπατε. Απλώς υπάρχουν δύο θέματα τα οποία μας ανησυχούν για τις ισοδονομίες. Καταρχήν, δυστυχώς τη στιγμή που προσπαθούμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά, χρειάζεται να προδικάσουμε ποιο θα είναι το μελλοντικό καθεστώς, γιατί αυτή τη στιγμή ε, πλανάτησε σε έναν αρκετά προβλέψιμο ορίζοντα που ξεκάθαρα θα το πω είναι αυτό του Brexit, το υπενθυμίσατε και εσείς ως εισηγητής και θυμόμαστε τι έγινε και με, με, την, 20, με την ισοδυναμία με τις ΗΠΑ. Είχαμε εκεί πρόβλημα με το Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε πως οι αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει στις κατεξουσιοδότηση πράτη στην ε, ισοδυναμία, στη φερεγγιότητα 2 δεν είναι το σύστημα το οποίο θέλει να προκρίνει η Κομισιόν. Όταν όμως ανακαλύπτουμε την τελευταία στιγμή και κατά τύχη και χωρίς διαφάνεια πως υπάρχει αυτό το σύστημα ισοδυναμίας, τότε δημιουργείται πρόβλημα και νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το πούμε απερίφραστα. Γιατί, επαναλαμβάνω, θα γίνει ακόμα πιο έντονο το θέμα αυτό στην, δυστυχώς ε, στα πλαίσια και του Brexit το οποίο εωρείται στον ορίζοντα. Ωραία. Πολύ ωραία. Δίνω το λόγο τώρα στην Κίη Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια που μας έκαναν γιατί ε, ξεκαθαρίζουν το τοπίο. Γιατί ακολουθήσαμε την λύση με τα εισοδήμανα Πρώτον, γιατί είχαμε την υποχρέωση εκπαίδευσης των παραγόγων, όπου ήμασταν πολύ πίσω από τη ΣΥΠΑ. Ε, γιατί τα δικά μας OTF καθυστέρησαν να εμφανιστούν, ενώ τα δικά τους CF ήταν ήδη στη θέση τους και για τα ισοδύναμα, ε, γι' αυτό το λόγο συζητούσαμε ε, τα ισοδύναμα στο σύστημα, για να μην χάσουμε όλη την εμπορική ροή από τους Ευρωπαίους επενδυτές που θα ε, μετακινεί το προς τη ΣΥΠΑ. Και για το κομμάτι το μετοχικό είχαμε πει για τις ε, με μετοχές της Apple που στην ε, Γερμανία είναι στο χρηματιστήριο ως ADR ε, το οποίο σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι επενδυτές είναι σε μειονεκτική θέση γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβαση στη βασική πηγή στην Αμερικανική αγορά. Αυτού του είδους συζητήσεις κάναμε και δεν ήταν οι συζητήσεις τόσο λεπτομερείς και το γεγονός ότι περνάμε τόσο χρόνο μετά την συμφωνία και όχι πριν, δείχνει ότι μπορεί στο μέλλον να ακολουθήσουμε άλλη τακτική και πως θα πρέπει η διαδικασία της ισοδυναμίας να μπαίνει στην αρχή της τριμερού, ε, του τριμερή διαλόγου και όχι να τον κολλάμε στο τέλος ως σύστατη λύση. Εσείς μιλήσατε για το παράδειγμα της Ελβετίας και θεωρώ πως υπάρχει μεγάλη διαφορά, τεράστια, από την δημιουργία ένα σύστημα ε, ε, ισοδυναμίας για διπλές εισαγμένες μετοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενό συστήματος όπου έχουμε δευτερογενή ε, συναλλαγή στο χρηματιστήριο όπου τουλάχιστον μία από τις μετοχές έχει μπει σε ε, χρηματογορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προηγουμένως treated them Όμως, εδώ η εταιρεία ισοδυναμία κατά Ελβετία δεν λαμβάνει υπόψη τη διάσταση αυτή που μόλις αναφέρατε και πρέπει επιγόντως να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε οι εκτός χρηματοστηριακές ε, ε, συναλλαγές ε, να ενταχθούν στο σύστημά μας με ένα, πλήρημα, με ένα πλήρες σύστημα ισοδυναμίας χωρίς καθυστερήσει, γιατί κάθε μέρα που περνάει η μόνη αλλακτική που μένει για τις εθνικές αρμόδιες αρχές είναι η εξαίρεση. έτσι ώστε να μπορεί ε, κάποια εθνική αγορά να λαμβάνει υπόψη και τις ελβετικές ισοδυναμίες και όχι μόνο τις ευρωπαϊκές. Έτσι ώστε ε, να βρούμε μια επίσημη λύση και να μην ε, μας ε, παρασύρει η πραγματικότητα προς μια λύση που δεν την επιθυμούμε. Και νομίζω ότι όταν έχουμε τέτοιου είδους διπλή εισαγωγή είναι σημαντικό αυτό να το παρακολουθήσουμε. Ε, επιτηρώντας και παρακολουθώντας τι γίνεται, ξέρετε κι εσείς πως η εφαρμογή της MIFID 2 ήταν η 3η Ιανουαρίου του 2018 και 17 από τα 28 κράτη-μέλη ακόμα δεν έχουν εντάξει πλήρως τη MIFID 2. Ε, στο Εθνικό Δίκαιο και δεν εφαρμόζουν τον κανονισμό από την 3η Ιανουαρίου και μετά, το οποίο σημαίνει το 50% των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τους δικούς μας κανόνες. Οπότε, αν θέλουμε να δούμε ποια είναι η ισοδυναμία άλλων δικαιοδικασιών στον κόσμο, τι να τους πούμε, ότι εμάς οι μισοί δεν συμμορφώνονται. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Οπότε αν δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κανόνε ισοδύναμη, τι να κάνουμε, να στείλουμε συστήματα και για τι τρίτε χώρε, Αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα και οι τρίτες χώρε δυσκολεύονται να το δεχτούν. Οπότε πιστεύω πω αυτέ οι πολιτικέ αποφάσει που βασίζονται σε τεχνική γνώση αλλά δεν αποτελούν ένα επίσημο σύστημα, είναι μια ιδιαίτερη δυσκολία και είχα πολλέ καταγγελίε από του Ελβετού, για παράδειγμα, για το γεγονό ότι αυτή η απόφαση είναι για ένα χρόνο, ενώ πιστεύω ότι θα είναι μόνιμη απόφαση. Και αυτό αποδεικνύουν ότι το ζήτημα αυτό είναι πολιτικής φύση και όχι τεχνικής. Και δεν ξέρω πώς θα τετραγωνίσουμε τον κύκλο παρά μόνο να ξαναξεκινήσουμε βασιζόμενοι σε ένα σύστημα ισοδυναμίας απόφαση με μια επίσημη διαδικασία και να μην το κάνουμε κατακαιρματισμένα σε κάθε κομμάτι της νομοθεσίας μας, αλλά να ξεκινήσουμε από την αρχή εκ νέου. Το χειρότερο για μένα είναι το τι θα γίνει μετά το Brexit πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε υψηλότατο επίπεδο. Η ειδοποίηση 30 ημερών ισοδυναμία για τι χρηματοπιστικέ αγορέ δεν θα λειτουργήσει και οι αποφάσει, οι ισοδυναμίε είναι ήδη πολιτικοποιημένε. Οπότε το να γίνεται κατά περίπτωση ε, αγορά αγορά-αναγορά δεν θα μα ικανοποιήσει ούτε για του επενδυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε για τα κράτη-μέλη, ούτε για τα πρώην κράτη-μέλη που θα είναι πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε η ισοδυναμία είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και το αναγνώρισε ο Λόρτ Χέιλ, πρώην Επίτροπος, ότι δεν λειτουργούσε σωστά και πως χρειάζεται μια οριζόντια νομοθεσία για την ισοδυναμία και αυτό το έκανε βέβαια πριν το δημοψήφισμα για τον Brexit, οπότε καταλαβαίνω απόλυτα πως η κατάσταση έχει αλλάξει, αλλά θα έλεγα πως επήγει πολύ περισσότερο από ότι ποτέ να γίνει αυτή η νομοθεσία, έτσι ώστε οι κεφαλογορές Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι γνωστές ε, και φημισμένες σε όλη ε, την Ιφίλιο και να μην καταστραφεί η φήμη τους λόγω αυτών των πολιτικοποιημένων αποφάσεων που θα ε, κληθούμε να πάρουμε. Καρολίν, για τους φιλελεύθερους. Όχι, άρα λοιπόν catch the eye. Ashley. Well, thank you, President. Ήρθα σε αυτή την ελεγκτική συνεδρίαση για να δούμε και για τα τελωνία. Α, ζητώ συγγνώμη, αλλά ο πρόεδρο χρειάστηκε να αλλάξει τη σειρά. Έπρεπε να φύγει για το πίεση του. Γι' αυτό πέσατε στο Μίφιτ. Ναι, το κατάλαβα. Απλά θέλω να ξέρω πότε ενημερώσατε, γιατί εγώ το έλαβα στις 9 και 4 και ότι έπρεπε να έρθω για να συμβάλλω σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω στο χτεσινό mail. Ναι, αλλά τι ώρα. Anyway, it hadn't reached my office and my diary by the time. Κοιτάξτε, εγώ μόλις έφτασα στο γραφείο στις 9, δεν το είχα και μέχρι στις 9 και 45 δεν το είχα πάρει. Ε, Όμω τέτοιε τέτοιες αποφάσεις, εγώ πιστεύω θα πρέπει να ε, ε, διαβιβάζονται, γιατί παίρνουμε ένα σωρό email. Πάντως αυτό εξηγεί την απουσία μου, Πρόεδρε. Ε, λυπούμε. Θα ζητήσω από τις υπηρεσίες μας να ρωτήσουν, να ελέγξουν. Συγγνώμη πότε στάλθηξαν αυτά τα mail. Κάνε ένας άλλος για το MIFID 2. Oh, it was already sent uh, yesterday morning, before 12 o'clock, 11 o'clock and 38 minutes. Ε, νομίζω 11 και 38 στάλει εχθές. Λοιπόν, για κοιτάξτε τα συστήματα mail σας. Ωραία, τότε τελειώσαμε και με την ίδια σειρά ο κύριος Λούντερ και μετά ο κύριος Άσλεμαν. Κύριος Λούντερ. Uh, for the opportunity uh, uh, Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και για τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις που ε, υποβλήθηκαν. Καταρχά για τα παράγωγα. Να σας πω ότι η κάλυψη στα παράγωγα είναι εξαιρετικά ισχυρή γιατί έχουμε μόνο μία αντιστοιχεία με τη ε, ε, USC-AFTC. Ωστόσο αυτή η απόφαση αντιστοιχείας καλύπτει το 95% των swaps που συναλλάζονται εκτός ένωσης. Ε, παρακαλώ να ζητήσω τους συναδέλφους να πάψουν να συζητούν γύρω μου. Λοιπόν, υπάρχουν δύο κύρια κέντρα συναλλαγών. Η μία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ένα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο είναι η ΕΠΑ. Με την απόφαση CFTC για τη ΣΥΠΑ καλύπτουμε πάνω από το 95% όλων των επιτοκίων, των επιτοκίων εκτός Ένωσης. Έχουμε ακόμα μερικέ συναλλαγές με Σιγκαπούρη και Χογκόγκ. Δεν έχουν ακόμα υποχρέωση και ε, θα τους αναγνωρίσουμε μόλις θα θεσπίσουν τέτοια υποχρέωση εμπορίας, αλλά ε, εκεί μιλάμε για μονοψήφια ποσοστά. 1% το πολύ στις περισσότερες περιπτώσεις. Οπότε το θέμα είναι ότι μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικές αντιστοιχίες υπέρ των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων εάν η, χώρα έχει υποχρέω... η άλλη χώρα έχει υποχρέωση και άρα είναι υποχρεωμένη να μας αναγνωρίσει εμάς για κάποιο παράγο γιατί είναι αμοιβαία ρύθμιση πρέπει και εκείνοι να μας αναγνωρίσουν και άρα πρέπει να περιμένουμε μέχρι ότου θεσπιστεί μια τέτοια υποχρέωση εμπορίας. Πιστεύουμε όμως ότι το 2018 μάλλον θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις με τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ. Επόμενο σημείο για τη ΣΥΠΑ και την συμπερίληψη εναλλακτικών συστημάτων εμπορίας. Εάν κάνουμε την αντιστοιχία και αν κάνουμε σοβαρά την αντιστοιχία, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το σύστημα των τρίτων χωρών στο σύνολό του, εφόσον τώρα τα αναγνωρίζουμε και νομίζω πως αυτό το έχουμε επιτύχει. Δεν είναι δίκαιο να λέει κανείς ότι δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Έχουμε εξαιρετική ομάδα, έχουμε input από τις τρίτες χώρες βεβαίως, αλλά είναι αλήθεια πως αυτά τα συστήματα δεν μπορεί να είναι ε, απεικόνηση του δικού μας συστήματος. Ε, ε, μιλάμε για πολύ εξελιγμένες δικαιοδοσίες, όπως είπα, όπου έχουν ένα εξαιρετικά διαφανές και ανοιχτό σύστημα, το οποίο δεν ε, είναι ακριβώς το ίδιο σε όλες τις πτυχές με το σύστημα MIFID αλλά πάντως ε, αν ε, θέλουμε να δούμε αν έχουμε την καλύτερη εκτέλεση και ανταγωνιστικές τιμές μπορεί να σταθεί η στάξια στο ευρωπαϊκό. Και αυτό γίνεται στη ΣΥΠΑ. Έχω και κάποιες άλλες στατιστικές που αποδεικνύουν ότι κάνουμε την καλή, καλή σωστή δουλειά Έχουμε λοιπόν για τις μετοχές που υπόκειται σε αυτή την απόφαση ε, δέκα ευρωπαϊκές, και, και τέσσερις ε, ε, μετοχές EA ε, που μπορούμε να δούμε ποια είναι, ποιες είναι οι τιμές. Με χαρά μπορώ να σας πω ότι όλες οι μετοχές πάνε στο στενότερο τίκ, δηλαδή εκτελούνται σε, σε πένες. Μόνο μία εξαίρεση υπάρχει. Είναι ένας ε, εκδότης ο οποίος ε, ε, εκμεταλλεύεται το πιλωτικό τικ που εκτελεί σε πέντε πένες. Όπως είπαμε, στην εκτίμηση ε, αντιστοιχίας αναγνωρίζουμε το καλύτερο δυνατό ποσοστό εκτέλεσης ε, που υπάρχει σε, όλε σε όλες τις ΣΥΠΑ. Και σίγουρα δεν έχουμε λάβει ε, λάθος αυτή την απόφαση, ωστόσο ε, ούτως ή άλλως την παρακολουθούμε ε, και θα παρακολουθούμε ορισμένα ATS Μόνο εκείνα δηλαδή που κάνουν εμπόριο ε, ε, μετοχών. Είμαστε πεπισμένοι ότι λάβαμε τη σωστή απόφαση γιατί πρόκειται για πλατφόρμες εξαιρετικά διαφανείς και έχουμε το καλύτερο δυνατό ποσοστό εκτέλεσης ε, στις ΕΠΑ. Τώρα, για τις ΕΠΑ και τα μεγέθη ΤΙΚ, αυτό είναι θέμα για μας και για την ανταγωνιστικότητά μας και πιστεύω πως φέτος θα έχουμε ένα καλό σημείο εκκίνησης έτσι ώστε όταν θα ανανεωθεί αυτή η απόφαση να υπάρχει ευθυγράμμιση των μεγεθών τι ανάμεσα στην Ένωση και της, ε, την Ελβετία ώστε να μην, είμαστε, να μην είναι σε μειονεκτική θέση η ελβετική πλατφόρμα. Τώρα, από το Δεκέμβριο του 2017 έχουμε ε, τονίσει ε, την ρυθμιστική συνεργασία μετά την αναγνώριση για να παρακολουθούμε δηλαδή μετά την έναρξη της συνεργασίας και της αναγνώρισης με τις τρίτες χώρες τι συμβαίνει Επίσης περισσότερα ε, MOUs θα πρέπει να έχουμε με τις χώρε χώρες για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Θα είναι ένα πολύ καλό συστατικό. Και τέλος το θέμα της ανοιχτής πρόσβασης, άρθρα 35 και 36. Όλοι ξέρουμε πως η ανοιχτή ε, πρόσβαση έχει ανασταλεί. Για τους επόμενους 30 μήνες δεν θα κινηθεί τίποτα. Έχουμε χρόνο λοιπόν για να εξετάσουμε αυτή την πολιτική όταν δηλαδή θα εκπνεύσουν οι ισχύουσες εξαιρέσεις. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ο κύριος Σα Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα αναφέρω το σημείο με την σειρά μιλήσατε για την υποχρέωση εμπορία παραγόγων και να υπάρχει επιλογή να σταματήσει αυτό σε πάρα πολύ γρήγορα. Ε, το επιχείρημα είναι ότι αν υπάρχουν τέτοια μέσα, αν υπάρξει απότομη πτώση ρευστότητα, ε, δεν μπορούν να βγουν offline γιατί αυτό απαιτεί αλλαγή των τεχνικών ε, προδιαγραφών και βέβαια η αλλαγή τη τεχνικής προδιαγραφή χρειάζεται χρόνο. Και βεβαίως το σκεπτικό είναι να έχουμε κάτι για να το κάνουμε αυτό κάπως πιο γρήγορα. Έχουμε λοιπόν στο ΕΜΗΡ 2-2 ε, ε, εκεί που υπάρχει η υποχρέωση της ε, καθάρισης κάτι ανάλογο βεβαίως δεν υπάρχει λόγος να γίνει το ίδιο και στην υποχρέωση εμπορίας. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν στις οθόνες ε, μια ε, πολύ χρωμή εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τα εθνικά καθεστώτα ε, που υπάρχει το θέμα της αμοιβαιότητας μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών, αλλά σε κάποια χώρα υπάρχει απαγόρευση του να υπάρχουν αυτές οι οθόνες και βέβαια να σκεφτούμε ότι με τον Brexit η μεγαλύτερη χρηματαγορά θα φύγει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εικόνα θα αλλάξει πολύ, οπότε αν ξαναδούμε το θέμα θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε πιο ενιαίους κανόνες. Τώρα σε καταστάσεις όπου το καθεστώς είναι πιθανώς το ρυθμιστικό καθεστώς πιο ελαφρύ σε κάποιες χώρες. Ένα παράδειγμα που σκέφτομαι είναι Εάν ε, κάποιος ε, εμπορεύεται για λογαριασμό του συνήθως έχει την εξαίρεση εκτός εάν μιλάμε για συναλλαγές υψηλής συχνότητες αλλά οι νομικοί μας λένε ότι ναι, αν βρίσκεται κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται άδεια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται, δεν είναι ιδεώδης αυτή η κατάσταση οπότε το θέμα του κατά πόσον βεβαίως θα αντέξει αυτό στις εξελίξεις, τις μελλοντικέ το αναφέρουμε, το υπονοούμε στην αρχική μας δήλωση. Δηλαδή, έχουμε τις υποχρεώσεις για τις μετοχές ε, ισοδυναμίας μετοχών και παραγόγων, αλλά δεν έχουμε τίποτα για την διαφάνεια, οπότε βρήκαμε κάποιον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά ε, και βεβαίως ε, ε, εμείς μπορούμε να δούμε το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν υπάρξει, παραδείγματο χάρη, ναι, κάποιο σπάσιμο της ρευστότητα στην Ελβετία, δεν μπορούμε να το λάβουμε υπόψη. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη προσέγγιση των ε, υποχρεώσεων αυτών των τρίτων χωρών. Και από την πλευρά των επενδυτικών εταιριών το σύστημα είναι αρκετά περίπλοκο. Έχουμε ένα συνδυασμό εθνικών αποφάσεων, προσωρινών εξαιρέσεων, διαφορετικά καθεστώτα ανάλογα με το αν απευθυνόμαστε σε, σε μικροεπενδυτές, σε επαγγελματίες επενδυτές και υπάρχει και μεγάλη διακριτική ευχαίρεια. Οπότε εμείς θα λέγαμε να το ξαναδούμε το θέμα κάπως ευρύτερα. Λίγο σύντομα για το μέγεθος ε, των ε, ΤΙΚ ε, νομίζω ότι κατ' ουσίαν αντέγραψαν αυτοί το ευρωπαϊκό καθεστώς επειδή έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα σε μεγαλύτερο αριθμό μεγορών έχουν καταλήξει σε ένα πιο ανταγωνιστικό μέγεθος αλλά δεν είναι και μονοδιάστατη η εικόνα μπορεί να συμβαίνει και το αντίστροφο και εκεί πέρα οι ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες έχουν λιγότερα παράπονα θα έλεγα αλλά συμφωνήσαμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε και βεβαίως ε, σκεφτόμαστε και να δούμε την σχετική τεχνική προδιαγραφή και να λάβουμε υπόψη ε, όντως ε, το που βρίσκεται κύριος η ρευστότητα. Μια τελική παρατήρηση που ήρθα σε επαφή με τα κράτη-μέλη τα τελευταία νούμερα είναι ότι 10 χώρες δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει την ΜΥΦΙΤ 2 δεν είναι και φοβερό αποτέλεσμα δεδομένου του ότι είναι σήμερα 25 Ιανουαρίου και πρέπει να ισχύει από τις 17. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε. Θα έχουμε κάτι να συζητήσουμε όταν θα συζητήσουμε και την ΜΥΦΙΤ 2. Πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο λοιπόν να δώσω την προεδρία στην Κέι Good morning, everybody, and apologies, I didn't know I was chairing this session until a few minutes ago, so um, I... Συγχωρείτε, καλημέρα. Δεν ήξερα θα προεδρεύσω μέχρι πριν από λίγα λεπτά, οπότε ζητώ την κατανόησή σας. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού. Έχουμε τον εισηγητή, τον Ραμόν Τρεμόζα, οπότε έχετε τον λόγο. Thank you very much, Madam Chair, dear colleagues. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Να σας πω πως χτες έγινε μια εξαιρετικά ε, καρποφόρο συζήτηση μεταξύ σκιωδών εισηγητών και πιστεύω πως μετά τη συμφωνία εκεί ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συμφωνήσαμε όχι μόνο συγκεκριμένη διατύπωση για τις τροπολογίες αλλά παράλληλα και το πνεύμα σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε για μια σειρά από ε, ζητήματα. Πρέπει να σας πω πως το 2013 που ήμουν πρώτος ηγητής για το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πως το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στον Ευρωπαίο πολίτη είναι ακριβώς η στεναρή συνένεση για να στείλουμε ένα απερίφραστο μήνυμα δημοκρατικής, δημοκρατικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζοντας πως η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έχει κάνει καλή δουλειά. Νομίζω ότι είμαστε όλοι ε, ενωμένοι στον ίδιο δρόμο προσπαθώντας να επιτύχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Εμείς είπαμε για παράδειγμα πως η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θα πρέπει, αν κριθεί απαραίτητο, να μετακινήσει πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς για να καταφέρει καλύτερα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Για την ονομασία εδώ να σας πω ότι είμαι ανοιχτό. και μπορώ να ξανασκεφτώ ε, και τις χώρες που μπορούν να κατανομαστούν και τα λοιπά γιατί το έχω πει και στο παρελθόν, θα πρέπει να κατανομάζουμε και τις εταιρείε οι οποίες έχουν, σε οποίες έχουν επιβληθεί, επιβληθεί πρόστιμα και εμείς είμαστε κοινοβούλιο, δεν είμαστε φόρουμ συζήτησης, οπότε πρέπει να βάζουμε τα χαρτιά μας στο τραπέζι. Γι' αυτό είπα, είμαι ανοιχτό με ευέλικτο τρόπο να ε, προσαρμοστώ γιατί είναι πάρα πολλέ τροπολογίε που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι το θέμα αυτό του κατονομασμού, το οποίο είναι ευαίσθητο επί τη ουσία. Για τον φορολογικό ανταγωνισμό, για τις τράπεζες, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια των διάφορων ερευνών έχουμε συμφωνήσει πολλά και πιστεύω πως το αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό. Και τέλος, πριν ακούσω τα δικά σας σχόλια, Χαίρομαι ιδιαίτερα που δίνουμε αυτή την αρμοδιότητα στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να υποβάλει μια ετήσια έκθεση έτσι ώστε οι εθνικές αρμόδιες ε, αρχές για τον ανταγωνισμό να πιεστούν κατά τη. Γιατί και εκεί υπάρχουν ανεξάρτητοι φορείς οι οποίοι θα πρέπει να μην επιβαρύνονται με πολιτικούς διορισμούς αλλά να κάνουν τη δουλειά του σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι γι' αυτό θα χαρώ πολύ να πετύχουμε συνένεση και όταν μιλάμε για ανταγωνισμό στις εναέριες μεταφορές και εκεί θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη. είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση χτες ε, εδώ μετά την Επιτροπή όπου μιλήσαμε για θέματα ανταγωνισμού στον κλάδο της αεροπλοείας και πρέπει να σας πω πως χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και τις ε, κοινή για παράδειγμα περιφέρειες Ευρώπης, νησιά, τα οποία θα πρέπει να εξυπηρετηθούν από τις ε, εταιρείε αερομεταφοράς. Θα σας ακούσω με χαρά και θα ξεκινήσουμε μετά από τα σχόλιά σας την όλη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των σοσιαλιστών πιστεύω... Α, πρώτα ο ΕΛΚ, ο Ζίγκριτ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Κιώδης δεν είναι διαθέσιμο σήμερα και μου ζήτησε να πάρω το λόγο εκ μέρους του, λέει ο κύριος Μουρεσάν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή για όσα έχει κάνει για το σχέδιο έκθεσης και για τις τροπολογίες, προσπαθώντας να πετύχει ένα συμβιβασμό. Καλή η συνάντηση των σχεδόν χτες και η ομάδα μας πήγε Πρέπει να συζητήσουμε ακόμα κάποιες από τις τελευταίες τροπολογίες. Θα το κάνει ο εισηγητής, θα επαναδιατυπώσει και νομίζω θα παρουσιάσει και ένα νέο συμβιβασμό για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή είναι σε κρεμότητα. Αναμφίβολα έχουμε ε, ακολουθήσει την κατάλληλη πορεία. Εμείς θεωρούμε πως η πολιτική των ανταγωνισμών δεν, είναι, δεν θα πρέπει να είναι θύμα πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέμα εμπειρογνωμόνων, είναι τεχνική πολιτική και βεβαίως έχει ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θα πρέπει να θεσπίσουμε εμείς το πλαίσιο αλλά το να κατονομάσουμε εταιρεία, στο να θέτουμε υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω αν είναι δικός μας ρόλος και γι' αυτό εμείς θέλουμε λιγότερη υποκειμενικότητα ως πολιτική ομάδα και είπαμε ας αφήσουμε την πολιτική ανταγωνισμού στην Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί κάνει τη δουλειά της με πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Δεύτερον, εσωτερική τραπεζική αγορά. Εκεί έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά με την ε, Τραπεζική Ένωση, με το ε, εγχειρίδιο, το ενιαίο εγχειρίδιο ε, ενιαίων κανόνων, με την ε, όλη πολιτική που χαράξαμε. Έχουν γίνει πάρα πολλά πρόσφατα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχουμε πραγματική τραπεζική ένωση αυτή τη στιγμή. Και τρίτον, Κοιτάμε τις έρευνες που γίνονται για τη σύσταση καρτέλ και εμείς γνωμοδοτούμε γενικότερα και για την κατάχρηση δεσπόζουσα θέσης ε, κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε εκτός δηλαδή από το καρτέλ είναι και αυτό θέμα στο οποίο, για το οποίο πρέπει να ενημερώνεται η Ευρώπη. Τέσσερα, η Γεωργία. Εκεί συνεργαζόμαστε πολύ καλά με τον εισηγητή Υπάρχουν κάποιοι γεωργικοί όροι οι οποίοι καλό είναι να οριστούν με τον κατάλληλο τρόπο εξ αρχής έτσι ώστε μετά να μπορέσουμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Για τη φορολογία. Θεωρούμε πως θα πρέπει να πληρώνονται εκεί που ασκήθηκε η οικονομική δραστηριότητα και όπου τα κέρδη ε, σημειώθηκαν. Και η, κατα... η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατομελών πρέπει να αυξηθεί και τα ελάχιστη, οι ελάχιστοι συντελεστέ για του εταιρικού η ε, εταιρικό φόρο νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αναφέρονται εδώ. Διαφθορά. Πιστεύουμε πως στις κρατικές προμήθειες η διαφθορά πολλές φορές στρεβλώνει σοβαρά τον ανταγωνισμό και θέλουμε σε αυτό να είμαστε σαφείς. Και βέβαια στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και πολλές φορές έχουμε και χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην διαδικασία κρατικών προμηθειών. Ε, τώρα βέβαια η δημιουργία της ε, Ευρωπαϊκής εισαγγελία θα βοηθήσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και το αναφέρουμε στην έκθεση τώρα. Χρονικά, χρονικός προσδιορισμός. Δεν υπάρχουν πολιτικοί στόχοι που να έχουν καταφέρει να βρούνε ποια θα πρέπει να είναι η καλή χρονική συσχέτιση μεταξύ ε, κίνησης έρευνας και αποτελεσμάτων αυτής. Εμείς θα πρέπει να λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συγχωρείτε, ε, τι πρέπει να κάνει, αλλά όχι να της λέμε συγκεκριμένη έρευνα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό θα ήταν παρεμβατικό. Τώρα για την Ελβετία Νομίζω ότι αυτά τα είπαμε. Για τις εναέρειες μεταφορές, ναι, θέλουμε ισότιμου κανόνες παιχνίδου και βεβαίω να προστατεύσουμε και τον Ευρωπαίο καταναλωτή, ο οποίος θα μπορεί να κάνει ενημερωμένο κατάλληλα την επιλογή που επιθυμεί. Πάντω, πάμε καλά και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά για τα όσα κάνατε. Όσο πιο πολύ η έκθεση αυτή ε, ακολουθεί το ρόλο που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πολιτική ανταγωνισμού, τόσο μεγαλύτερη επιρροή θα ασκήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τα χρονοδιαγράμματα, γιατί ο κάθε ένας έχει πέντε λεπτά. Και μετά στο Catch the Eye φτάνουμε στα δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, και... αλλά ευτυχώς ε, ε, μέσα στο χρόνο ήσασταν, αν και δεν ξέρατε πόσο χρόνο σας είχα δώσει. Επόμενος ο σκιώδης του Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Ε, έχουμε ένα καλό σύνολο τροπολογιών πιστεύω καθώς και μια καλή βάση εργασίας με τη βάση της συμβιβαστική που έφτιαξε ο εισηγητής. Και σημαντικοί τομείς αναγνωρίζονται τόσο το κείμενο του εισηγητή όσο και οι ε, τροπολογίε τροπολογίες. Ε, εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τον πιο αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα του ανταγωνισμού. Αυτό είναι ο στόχο των τροπολογιών. Οι τροπολογίε που αφορούν την Google επίση νομίζουμε ότι είναι σωστέ. Είναι κατανοητό να έχουμε την Google εδώ ως ε, ε, την αιστεία αυτού του τομέα και με σαφή τρόπο και λογικό γιατί δεν μπορούμε να το, αγνοήσουμε. Αν και συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι σε αυτό το θέμα, ενώ θα εξασφαλίσουμε ότι αντικατοπτρίζονται οι βασικές μας ανησυχίες στο τελικό σχέδιο. Για τον ψηφιακό τομέα, Έχουμε τις, ε, τους οργανισμούς online, έχουν κατατεθεί καταγγελίες και παραπάνω, ας πούμε, οι, οι εταιρείε ε, πολλές φορές ε, έχουν κατηγορηθεί ότι δεν δίνουν αρκετές πληροφορίες όταν κανείς προσπαθεί να κάνει ε, κρατήσεις θα πρέπει να έχουμε αρκεί νομοθετικά οχήματα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ευθυνότερες πτήσεις και πρόσβαση σε αυτές για την, τις ευρωπαϊκές πτήσεις. Κάτι ακόμα που πρέπει να τονιστεί είναι η εφιέρωση των ιδίων πόρων στην DG ανταγωνισμού. Νομίζω, συμφωνώ πως θα πρέπει να προσεχθεί αυτό το ζήτημα για να ανακατανεμηθούν οι πόροι της Ένωσης, όμως έχουμε υπογραμμίσει σε διάφορες τροπολογίες και σε δική μου ότι αυτό θα πρέπει να συμβαδίσει με την ε, διαδικασία διαφάνειας μεταξύ των όσων σχεδιάζουν τις κατευθυντήριες γραμμές και των όσων τις εφαρμόζουν. Ε, θα πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου η DG, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, να είναι και ο δικαστής και ε, η ένορκη και ε, ο μάρτυρας υπεράσπισης και ο μάρτυρας κατηγορίας. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να επιτύχουμε τους στόχος μας, αλλά όχι μόνο προς χάρη της απελευθέρωσης. Να είμαστε βέβαιοι ότι η υπηρεσία των βασικών οικονομικών συμφερόντων θα εξασφαλίζεται στις πιο προσιτές τιμές ολόκληρη την Ένωση και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις νησιωτικές και περιφερειακές οι πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ένωσης. Και αυτό είναι και το νόημα των τροπολογιών του εισηγητή. Όταν αναλύουμε τις επιλογές της παγκοσμιοποίησης, να εξασφαλίσουμε πως στήρουν τα κοινωνικά στάδια στάνταρ προς όφελος των όσων εργάζονται στον τομέα αλλά και προ όφελο των καταναλωτών και τέλος είμαι επίση ευτυχής ότι που διατηρούμε αυτή την πίεση τονίζουμε το θέμα της, ε, του ανταγωνισμού και στον τομέα της γεωργίας. Υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές ανάμεσα στις τιμές των τροφίμων που προφέρονται στον τελικό καταναλωτή και των τιμών που προσφέρονται στους γεωργούς για τα προϊόντα τους. Αυτό θα πρέπει να το χειριστούμε και στις τροπολογίες και στις συμβιβαστικές και να στηρίξουμε τη δράση που λαμβάνει υπόψη τους ε, παραγωγούς μικρής κλίμακας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να συμφωνήσω και εγώ με τους συναδέλφους του ΕΛΚ και των Σοσιαλδημοκρατών. Συγχαρώ τον Ραμόν Χτες ε, είδαμε κάποιες πολύ καλές ε, συμβαστικές ε, προτάσεις. Τώρα δεν θα σταθώ στη δουλειά του εισηγητή, αλλά στις τροπολογίες που ακόμα κυκλοφορούν, που καλύπτονται εν μέρη από τις συμβαστικές προτάσεις, εν μέρη όχι. Υπάρχουν τέσσερα ζητήματα. Πρώτον, θα ήθελα να τονίσω αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Μουρεσάν του ΕΛΚ. Πρέπει να είμαστε εστιασμένοι, να θυμόμαστε ότι είναι μια έκθεση για τον ανταγωνισμό, δεν θα πρέπει να αφορά τους φόρους, τις πληρωμές, ούτε να γίνει έκθεση για το Google, αν μου επιτρέπετε. Αλλά νομίζω ότι ο εισηγητής το έχει καταλάβει. Ε, ειδικά αν δούμε τις πρώτες συμβαστικές τροπολογίες, βλέπετε ότι τονίζει την σημασία του να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να μην υπάρχει επιλεκτικότητα στις ε, κρατικές ε, ενισχύσεις ναι, και εκτιμώ πράγματι το έργο σας. Από την άλλη βλέπω ότι υπάρχουν πολλές ε, τροπολογίες ε, μεμονωμένες ε, διαφόρων συναδέλφων που πηγαίνουν πέρα από το πεδίο εφαρμογής και αυτό ανισχύει την ομάδα μας για να είμαστε εστιασμένοι. Δεύτερον, όπως ανέφεραν, ανέφερε και ο συνάδελφος ο κ. αν πρέπει να σεβόμαστε την ανεξαρτησία τη Γενική Διεθνής Ανταγωνισμού. Ο καθένα έχει την δική του δουλειά και υπάρχει η Γενική Διεύθυνση η οποία είναι αρμόδια για την επιβολή τη πολιτική που εμεί χαράζουμε. Το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει κάποιε γενικέ παρατηρήσει για το πλαίσιο τη πολιτική, αλλά δεν θα πρέπει να κρίνουμε συγκεκριμένε περιπτώσει. Ε, γι' αυτό ακριβώ είμαστε και επιφυλακτικοί για το να κατονομάζουμε συγκεκριμένες χώρες ε, και κράτη-μέλη. Και ακριβώς προτιμάμε μια πιο γενική διατύπωση τρίτων. Ε, καλό είναι να σεβόμαστε ο ένα στην δουλειά του άλλου, ειδικά όταν μιλάμε για ανοιχτά θέματα. Βλέπω ότι ο εισηγητής έχει επίδειξει αυτόν τον σεβασμό δεν ε, μπαίνει σε πολλές λεπτομέρειες για τις ε, τρέχουσες εκθέσεις. Απ' την άλλη υπάρχουν πολλές τροπολογίες ακόμα που κατά την άποψή μου ε, πηγαίνουν πολύ μακριά για το 2 CTP, 3 CTP παραδείγματος χάρη, φορολογικά ζητήματα, πράγματα τα οποία είναι ανοιχτά για την, ή και για την κοινή εταιρική φορολογική βάση Και τέταρτο και τελευταίο, ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει περιληφθεί ναι, και νομίζω ότι πρέπει να το προσέξουμε αφορά ακριβώς ε, το θέμα αυτό του προγράμματος ε, αγορών ε, στοιχείων διαφόρων σε σχέση με τον ανταγωνισμό της εσωτερικής αγοράς. Βλέπουμε πως οι εθνικές κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να δικαιολογήσουν ε, επιλεκτικές αγορές εταιρικών ομολόγων. Ε, είχαμε μια συζήτηση με την κυρία Βεστάκερ, είχε πει την προηγούμενη φορά ότι θα το σκεφτεί και θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις και ενδιαφέρον θα ήταν νομίζω να υπενθυμίσουμε ε, τα δέσμευσή της στην κυρία Επίτροπο. Του τελευταίντος καλό είναι να συνεχίσουμε τις ε, επικοδομητικές συζητήσεις που ξεκίνησαν χθε. Ευχαριστώ, δεν βλέπω άλλον σκιωδή εισηγητή, οπότε όποιος άλλος θέλει μπορεί να μιλήσει. Η Περβάνα λοιπόν, για δύο λεπτά. Επιτρέψτε μου καταρχήν να καλωσορίσω μία ομάδα ακροατών, είναι δημοσιογράφοι, ε, που έχουν έρθει για ένα ε, σεμινάριο στην Ακαδημία η Ευρώπη μας Jacques Delors και να ξεκινήσω λέγοντας πως δεν βλέπω τη δυνατότητα συμβιβασμού και επανέρχομαι στις τροπολογίες που έχω καταθέσει πιστεύω πως είναι σημαντικό να τις βρούμε μέσα στο συμβιβασμό και ξεκινώ με μια γενική παρατήρηση για αυτή την έκθεση, την ετήσια έκθεση. Βεβαίως δεν μπορούμε να μπούμε κατά περίπτωση ε, σε θέματα υποθέσεων ανταγωνισμού που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο στον ορισμό του γενικού πλαισίου επεμβαίνουμε και σε μια ετήσια έκθεση δεν μπορούμε όμως να μην κάνουμε καμία αξιολόγηση υποθέσεων οι οποίες έχουν κλείσει, έχουν ληφθεί από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μου φαίνεται γκροτέσκο κάτι τέτοιο και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτό τον όρο. Για την Google και την Apple, ολόκληρο ο πλανήτης έχει σχολιάσει τι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο εμεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Είναι αυτό ορθή πρακτική. Αντίθετα, στην ετήσια έκθεση έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία σφαιρική και συγκεκριμένη ανάλυση των αποφάσεων που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και προς αυτή την κατεύθυνση υπέβαλα ε, τις τροπολογίες, για παράδειγμα, για την έρευνα που τρέχει αυτή τη στιγμή για τις ε, συνθήκες εκμετάλλευσης ε, ε, των όσων εργάζονται στα McDonald's ή την επίπτωση που θα έχει η συγχώνευση Monsanto-Bayer, γιατί είναι νόμιμες αυτές οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου και καλό είναι να αναφέρονται. Και στο τελευταίο σημείο, για να μην ξεπεράσω το χρόνο μου, έχουμε μια σειρά τροπολογιών τις οποίες κατέθεσα για τις διεθνείς επιπτώσεις της δικής μας πολιτικής ανταγωνισμού, γιατί πιστεύω πως ο συσχετισμός μεταξύ της δράσης Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και του διεθνούς εμπορίου είναι ένα σημείο στο οποίο χρειάζεται να κάνουμε πρόοδο. Και αυτό βέβαια με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλος κανείς για το Catch the Eye? Κύριε Λάιτενμπεργκερ, σας καλωσορίζω και αν θέλετε να ε, κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο, με χαρά θα σας ακούσω. Αξιότιμα μέλη, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέψετε... Καλωσορίζουμε ε, και την παρακολούθηση των θεμάτων μας που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα σχόλια που έχετε υποβάλει στα πλαίσια της εκθεσής σας και να σας πω πως για την Επίτροπό μας και πραγματικά εκτιμάμε ιδιαίτερα ε, τον επικοδομητικό διάλογο που κάνουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως επίσης και τα όσα συζητάμε εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τους χειώδεις εισηγητές, θα τα συζητήσουμε θα κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά ό,τι έχετε ε, βάλει στο ψήφισμα και θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες. Τώρα θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ε, παρατήρηση ε, για το πόσο είναι εμπρόθεσμη και αποτελεσματική η, επιβολή των αποφάσεων είναι ένα στοιχείο που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Και είναι ένα θέμα το οποίο και η Επίτροπος θέλει να λάβουμε υπόψη στον εξυγχρονισμό των εργοσιών. There is not a single um, measure that unties the Gordian ε, να σας πω πως δεν μπορούμε να αφήσουμε το θέμα της διάρκειας των ερευνών εκτός πεδίου συζήτησης. Πρέπει να έχουμε στοχευμένα ερευνητικά εργαλεία, να μπορούμε να τελειοποιήσουμε την πρόσβαση, για παράδειγμα, στους φακέλους των επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό έρευνα, να δούμε τι γίνεται ε, με τη δημιουργία ε, δωματίων για εξέταση απόρριτων εγγράφων και βεβαίως να συνεργαστούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία μαζί σας και να δούμε τι γίνεται και με τα θέματα διακανονισμού σε καρτέλ και με τις υποθέσεις αντιτράστ ε, και πώς μπορούμε εκεί να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Η επιβολή αποφάσεων αντιτράστ έχει να κάνει με την εταιρική συμπεριφορά, η οποία είναι βλαβερή και η οποία χρειάζεται να απαγορευτεί και επίσης να τιμωρηθεί. Πολλές φορές πρέπει να είμαστε επεμβατικοί και η νομολογία τονίζει την ανάγκη ε, να είναι πολύ σαφή ε, τα ευρήματά μας και αυτή τη στιγμή την ομολογία το δίδαγμα είναι πως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο θέμα αυτό της ακρίβειας των δεδομένων που παρουσιάζουμε. Οπότε όταν κοιτάμε τους τρόπους και τη μέθοδο για να επιταχύνουμε τις υποθέσεις δεν θα πρέπει να πιστεύουμε υπερβολικά πολύ με μονομένα στοιχεία όπως ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα γιατί μπορεί να χρειαστούν παραπάνω συζητήσει για να δούμε ποια είναι η σχέση κόστους ωφέλους αυτών. Και τελικά να δούμε ότι κάτι άλλο είναι πιο σημαντικό από το να τρέξουμε να προλάβουμε κάποιο, κάποια προθεσμία. Χαίρομαι που μιλήσατε για τους οικονομικούς και τους ανθρώπινους και τους τεχνικούς πόρους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στην αγορά και εκτός αυτής. Και το big data και η τεχνητή νοημοσύνη, τα μεταδεδομένα δηλαδή και η τεχνητή νοημοσύνη είναι τα θέματα που μας απασχολούν. 5-2 terabyte ε, δεδομένων η Google. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί πρέπει να το κοιτάξουμε και συστήνω σε εσά συνιστώ σε εσά και στην ε, Επιτροπή σας να παρακολουθήσετε στη συζήτηση για προοπτικές ε, της Ευρωπαϊκής, χρηματοδοτικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα έτσι ώστε να μας πρικοδοτήσετε με τους απαραίτητους πόρους για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Το αφήνω εδώ. Υπάρχει μια σειρά από συγκεκριμένα θέματα που έχουν τεθεί. Συνάδελφοι και εγώ είμαστε στη διάθεσή σας. Για να τα συζητήσουμε, για να σας ενημερώσουμε και θα ήθελα να προχωρήσει ο διάλογος ε, με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο. Και σας ευχαριστώ για τα επικοδομητικά και ορθά σας σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή χαίρεται που σας είχε μαζί και χαίρεται για τη δέσμευση ε, και τη συστράτευση που δείχνει η δική σας ομάδα και τον τρόπο που εξηγείτε τη δουλειά σας σε όλα τα μέλη του Βουλίου. Στρέφουμε ε, προς τον εισηγητή για καταληκτικά σχόλια. Ένα λεπτό. Ραμόν. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Βεβαίως είμαι στην διάθεσή σας για να ξαναγράψουμε αν θέλετε συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Ξέρετε πως υπάρχουν πολλές τέτοιες για... από πολλούς βουλευτές και προσπαθούμε να τα προσαρμόσουμε. Αν δεν συμφωνούμε σε κάποια πράγματα θα τεθούν σε ψηφοφορία. Αλλά πάντα εγώ θέλω να υπάρχει ε, ευρεία συνένεση κυρίως ε, γιατί έτσι μπορούμε ακριβώς να δώσουμε ένα μήνυμα και μια δημοκρατική εντολή προς την ε, Κομισιόν τη διαπραγματευτική ομάδα και βεβαίως τους πολίτες μας. Για τα άλλα θέματα αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν θέλουν να μπουν τόσα πολλά θέματα φορολογίας, αλλά στην περίπτωση κάποιων εταιριών υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Η Google, παραδείγματος χάρη, αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2013. και βεβαίως ε, η Google έχει αυξήσει ε, το μερίδιο αγοράς από 50% σε 95% σε πολλές χώρες στην Ευρώπη και κατέστρεψε πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες. Άνθρωποι από πολλές χώρες ε, ήθελαν ακριβώς να ερευνήσει η Κομισιόν το θέμα αυτό. Αυτά είναι γεγονότα και όταν πάω στη χώρα μου δηλαδή με ρωτά ο κόσμος «Ε, τι κάνετε στο κοινοβούλιο και λέμε γράφουμε περιπτώσεις ε, γράφουμε εκθέσεις για περιπτώσεις που απασχολούν τον τύπο που είναι σοβαρά πράγματα δεν μπορούμε να παριστάνουμε ότι είμαστε σε συνθήκες εργαστηρίου και αυτό ακριβώς ε, εγώ θέλω να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα. Θα τα ξαναπούμε στο Στρασβούργο. Και ελπίζω να έχουμε την απαραίτητη συνένεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους όσους μίλησαν. Αντιλαμβάνομαι ότι ήδη βρίσκεστε στις συζητήσεις με τους κοιόδης ε, για το χρονοδιάγραμμα να σας πω ότι ο στόχος θα είναι να πάμε σε ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 21 Φεβρουαρίου και αργότερα βεβαίως στην ε, Ολομέλεια. Λοιπόν, Ελπίζω να έχετε ολοκληρώσει μέχρι 21 Φεβρουαρίου. Ε, είμαστε και μπροστά από το πρόγραμμα. Δεν σημαίνει συχνά. Αυτό σημαίνει όμως ότι έχει έρθει εδώ συγητής για το επόμενο θέμα. Αλλά να δω ποιος άλλος έχει έρθει. Επειδή υπάρχουν οι από τις μεγάλες ομάδες, ε, και ο εισηγητής ε, ε και 44 είναι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Ρομπετσίλη από το ECR. Έχετε τον λόγο. Ε, ευχαριστώ και οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας μας, συνεισφέρει στην ανάπτυξη Και βεβαίως ε, δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι και θέμα τεχνολογίας ε, και άλλων ζητημάτων. Βεβαίως από την άλλη κάποιες επενδύσεις έχουν ε, κίνδυνο όχι τόσο για τη χώρα η οποία τις δέχεται, αλλά για άλλες γειτονικές που μπορεί να ε, φύγουν. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο για να εκφράσουν ακριβώς ανησυχίε τους στι γειτονικές χώρες. Υπάρχουν λοιπόν τώρα ένα σύστημα εξέτασης ε, των επενδύσεων αυτών και το επίπεδο βεβαίω ποικίλει από χώρα σε χώρα και η πρόταση της Κομισιόν είναι μια πρόταση ταχεία εξέτασης ε, και θα έχουμε έτσι και πληροφορίες που θα συλλέγονται από τους χρήστες και οπωσδήποτε αν ακούσατε και τον αρμόδιο επίτροπο θα ακούσατε ότι πάντα φέρνει ως παράδειγμα την ε, Κίνα και προς τα εκεί πηγαίνει αυτή η πρόταση. Γι' αυτό λοιπόν έχω κάνει κάποιες ε, προτάσεις για να αλλάξει αυτή η έκθεση και θα προσπαθήσω ακριβώς να εξηγήσω τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε τα ζητήματα ασφάλειας και δημόσιας ε, τάξης. Ε, ο ορισμός ε, μπορεί να γίνει πιο πολυπλοκός βεβαίως όπως παραδείγματος χάρη να, να μιλάμε για έμεσες ξένες επενδύσεις υπάρχουν κάποιοι ορισμοί που βλέπετε στην έκθεσή μου γιατί μπορεί να κάποιες εταιρείε ή φυσικά πρόσωπα να το κάνουν μέσω ενός άλλου κράτους μέλους μέσω ενδιάμεσου δηλαδή γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να περιληφθούν και αυτές οι περιπτώσεις στον έλεγχο οπότε για να καλύψουμε και άλλες επενδύσεις ε, τρίτων χωρών Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ο εισηγητής ε, πιστεύει ότι τα σημεία αυτά επαφής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσει η Κομισιόν πληροφορίες για το ποιος είναι τελικά ο επενδυτής ε, και οι χώρες ε, που επενδύουν σε άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες με τον καλύτερο τρόπο και από τα κράτη-μέλη μέσω υποβολής ε, πληροφοριών όπως προτείνεται ε, σε ένα σημαντικό ζήτημα θέλουμε να περιληφθούν και τα μήνυε στις κρίσιμες υποδομές γιατί η δημόσια τάξη πλέον εξαρτάται από την ιδιοκτησία των μήνυε και βλέπουμε ότι αν είναι σε χέρια ξένων μπορεί να υπάρξουν διάφορα σημαντικά ζητήματα. Επίσης επεκτείναμε και την γεωγραφική κάλυψη, καλύπτονται και τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών γιατί υπάρχουν επενδύσεις και εκεί και έχει και αυτό γεωπολιτική σημασία. Περιλάβαμε επίσης και τον αριθμό των, και τους φορολογικούς παραδείσους, ο αριθμός των οποίων μειώθηκε πρόσφατα, αλλά ξέρετε ότι και από εκεί διοχετεύονται ξένες επενδύσεις στα κράτη-μέλη. Μετά έχουμε και επενδύσεις χαρτοφυλακίου, εάν είναι ιδιαίτερο σημαντικές για κάποιο κράτος μέλος. Και βεβαίως ένα άλλο επίμαχο ζήτημα είναι Ε, επενδύσεις ε, για αμυντικούς ε, σκοπούς που δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε επιπλέον έλεγχο. Γιατί γιατί το να επενδύει ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ σε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δημιουργεί κίνδυνο, δημιουργεί περισσότερη ασφάλεια αν μιλάμε για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ξέρω πως είναι ευαίσθητο πολιτικά το ζήτημα, απλά το ανοίγω εγώ και θα ήθελα να το συζητήσω με τους συναδέλφους για να βρούμε την καλύτερη λύση. Η εμπιστευτικότητα. Και εκεί θα θέλαμε να υπάρχει κάποια εμπιστευτικότητα των πληροφοριών γιατί είναι ευαίσθητες πληροφορίες, δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι αρχές, αλλά έχει μεγάλη σημασία η εμπιστευτικότητα. Συμπερασματικά. Θεωρώ ότι το σύστημα αυτό ελέγχου δεν θα σταματήσει τις άμεσες ε, ξένες επενδύσεις ε, γιατί γνωρίζουμε ότι λίγες είναι αυτές και έχουμε σε άλλα κράτη-μέλη συσσωρευμένο πλούτο. Γι' αυτό είναι ευκαιρία έμεση ξένες επενδύσεις ε, για κάποια κράτη-μέλη να έρθουν πιο κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στους Σκιώδη Εκ μέρου του ΕΛΚ, παρακαλώ, είστε η πρώτη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία την οποία μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ακολουθεί την ε, κατάλληλη κατεύθυνση και μπορούμε να θεωρήσουμε ως ένα πρώτο στάδιο. Επίσης οι άμεσες ε, ξένες ε, επενδύσεις είναι απαραίτητες. Δεν υπάρχει θέμα, είναι απαραίτητες για την Ευρώπη και για τα κράτη-μέλη και να σας πω πως είμαστε μίες από τις πρώτες ε, γεωγραφικές ε, ζώνες στον κόσμο στον οποίο επενδύονται ξένα κεφάλαια και θα πρέπει να παραμείνουμε στην κορυφή αυτού του καταλόγου γιατί για την απασχόληση στην Ευρώπη, στα κράτη-μέλη, τα όσα διακυβεύονται είναι πάρα πολλά. Αυτά και παράλληλα θα πρέπει να παραμείνουμε λογικοί, όχι αφελείς, να ευαισθητοποιηθούμε και να ξέρουμε πως η Ευρώπη έχει τεχνολογία, έχει γνώσεις που είναι μοναδικές και που είναι ε, ε, εχμής σε πολλούς στρατηγικούς ή όχι κλάδους και μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν ορέξεις. Το σύστημα φιλτραρίσματος, screening των επενδύσεων είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι καλοδεχούμενο για να προστατεύσει τις υποδομές μας, την τεχνολογία μας, την κυριαρχία μας και βεβαίως την ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης, το οποίο είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις, κάποιες προτάσεις για συγκεκριμένα σημεία. Να σας πω καταρχήν πως κρίνω σημαντικό να μην περιορίσουμε το screening στις στρατηγικές επενδύσεις, αλλά να καλύψουμε να είμαστε πολύ ανοιχτοί και όλες τις υπόλοιπες, λαμβάνοντας υπόψη ποιο είναι το σύνολο των επενδύσεων το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είναι ευαίσθητο το να ε, αποκλείσουμε κάποιες παρόλο που δεν υπάρχει ε, συγκεκριμένη αναλογικότητα μεταξύ της ε, επιρροής όσους έχουν μετοχών επιχειρήσεων και των επενδυτικών ποσών που καταθέτουν γιατί πολλές φορές είναι μια ελάχιστη συμμετοχή που μπορεί αυτή τελικά να επηρεάσει σημαντικά και να αποτελεί μόνο μια πρώτο, ένα πρώτο στάδιο. Οπότε να μην τους αποκλείσουμε. Για τη διάκριση που προτείνεται στο screening μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών τρίτων χωρών θεωρώ πως είναι θέμα προσυζήτηση. συζήτηση προσωπικά είμαι μάλλον υπέρ της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας αφήνει την δυνατότητα να κάνουμε ένα screening όλων των επενδυτών από όπου και να προέρχονται που είναι αυτό το οποίο γίνεται νομίζω έτσι και αλλιώ στο σύνολο των χωρών ε, για το σύνολο των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μίντια και τις υποδομές τις κρίσιμες υποδομές θεωρώ πως είναι μια καλή πρόταση και πως θα έπρεπε να πάμε και λίγο παρακάτω αεροναυπηγική και αερομεταφορές και για την ανάγκη διαδικασιών που θα είναι ταχύτατες θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναλύσουν την κατάσταση μέσα σε πολύ σύντομες προθεσμίες και θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη που υπάρχει για συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Είδαμε πως έγινε μια ακρόαση στην αρχή της εβδομάδας και η Επίτροπος μας υπενθύμησε πόσο δύσκολο είναι να συλλέξουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν για το τι γίνεται ή όχι στα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κληθούν να παίξουν το παιχνίδι, αλλά βέβαια χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο εμπιστευτικότητας για όλες αυτές τις πληροφορίες. Νομίζω μπορούμε να το πετύχουμε. Χαίρομαι που μπόρεσα να μιλήσω για τα σημεία αυτά με τον εισηγητή και τους σκιώδες. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που ε, σεβαστήκατε την χρονοθυρίδα σας σήμερα το πρωί. Το, μας δίνει ένα περιθώριο ο κύριος Ήβαν για τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ. Η δική μου παρέμβαση θα είναι συντομότερη. Είναι προφανές ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν πολύ σημαντικό ρόλο για την ευρωπαϊκή οικονομία και δεν μιλώ μόνο για την απασχόληση αλλά και για τη μεταφορά τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, πολλά, για τους δεσμούς που μπορεί να δημιουργηθούν ανάμεσα στο, ε, στις οικονομίες ε, και στην... Ε, μπορούσε έτσι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για να παληθεύει, να ελέγχει τις επενδύσεις αυτές οι Κομισιόν, γιατί όλες οι άμεσες επενδύσεις δεν έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, δεν έχουν πάντοτε θετικό αντίκτυπο δε για το ευρωπαϊκό project εν γέννη. Υπάρχουν παραδείγματα που αυτές οι επενδύσεις έρχονται και θέτουν ακόμα και σε κίνδυνο το ε, τα ευρωπαϊκά project. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τη χώρα προέλευσης ε, των επενδύσεων αυτών. Όλες οι χώρες που βρίσκονται στον κατάλογο των ε, χωρών που είναι παράδειση φορολογική και τα θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό Ευρωπαϊκή Ένωση να ανορίζει ποια είναι η επιρροή αυτών των επενδύσεων τελικά. Να μπορούμε δηλαδή να υπολογίσουμε ε, τις συνέπειες, γι' αυτό και ε, θα ήθελα ε, να συνεχίσουμε τις εργασίες. Για την ώρα αυτά έχω να σας πω. Δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον οπτικού εδώ. Άλτε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το σχέδιο έκθεσης ε, καταρχάς των εισηγητή. Ε, περιλαμβάνονται εδώ πολλές ιδέες που ενισχύουν ε, την ευρωπαϊκή πρόταση. Για παράδειγμα, καλωσορίζω την επέκταση του πεδίου για επενδυτέ τρίτης, ε, τρίτων χωρών. Ε, εν γέννη, ε, οι άμεσες καίνε επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές γιατί φέρνουν θέσεις απασχόλησης Είμαστε ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στον κόσμο και θα πρέπει στους επενδυτές να προσφέρουμε ε, διαφάνεια. Όπως είπε όμως και ο πρόεδρος Γιούνκερ, δεν είμαστε και αγαθοί και ανόητοι. Ε, η Ευρώπη πάντοτε πρέπει να υπερασπίζει τα στρατηγικά της συμφέροντα. Ε, και αυτό αναμένουν οι πολίτες της Ένωσης. Με χαρά βλέπω την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό. Αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν διαβλέπει την αξία μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε σχέση με το σ άμεσες ξένες επενδύσεις και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή αν σκοπεύει να δίνει μόνο ε, ε, πληροφορίες σε σχέση με την ε, τα οικονομικά ζητήματα. Ο, ο συμβουλευτικός ρόλος σας επιτρέπει να προστατεύετε τα συμφέροντα της Ένωσης και εγώ ως κοιόδης εισηγητής θα ήθελα να σας δώσω μια πρόταση που μας επιτρέπει συλλογικά να απαντήσουμε και να υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα όταν αυτά κινδυνεύουν. Για παράδειγμα, θα είχαμε πουλήσει το ελληνικό λιμάνι στη, χωρίς την δημοσιονομική κρίση και θα το είχαμε αυτό συνδέσει με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα ήθελα αυτά τα ζητήματα να τα εξετάσουμε από κοινού με τους, τον εισηγητή και τους συναδέλφους. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω το σκιώδη εδώ των πρασίνων. Ναι, εγώ αντικαθιστώ τον Έρνεστ. Ευχαριστώ με την έκθεση κύριε Ζήλε για την καλή βάση που μας δώσατε και γιατί διευκολύνεται αυτή τη συζήτηση για την πρόταση της Κομισιόν που εν γέννη είναι πρόσδεκτη. Βασικός στόχος της πρότασης είναι η διευκρίνηση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης Θέλουμε λοιπόν να επαληθεύσουμε την ισχύ αυτής της πρότασης. Στο άρθρο 4 η Κομισιόν διευκολύνει την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη και συνδέει σε αυτά οικονομικά κριτήρια. Αυτή η έννοια καλύπτει και το κατά πόσο έχουμε να κάνουμε με ε, κυβερνήσεις συγκεκριμένε έχουμε να κάνουμε και με τα θέματα ασφάλειας, κρίσιμη σημασίας ε, ή εθνικής σημασίας. Πρέπει επίσης να συζητήσουμε και το θέμα των άμεσων επενδύσεων. Επίσης προτείνεται εναρμόνιση, στοιχεία εναρμόνισης, προτείνει μηχανισμούς ελέγχου στα κράτη-μέλη, διαφάνεια, όχι έλλειψη διακρίσεων και πληροφορίες σε σχέση με την οικονομική κατάσταση του επενδυτή. Ε, θέλουμε να κάνουμε μια πιο συνεπή ε, βιομηχανική πολιτική προστίθεται μια νέα διάσταση Επίσης, αυτό το όργανο συμβάλλει στη βελτίωση του συντονισμού και της συνεπούς δράσεις απέναντι σε τρίτους εταίρους κλειδιά, ειδικά αυτούς με τους οποίους έχουμε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις ήδη. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια πιο συνεπή ε, δράση σε σχέση με τις εξωτερικές μας σχέσεις και όσον αφορά την πρόταση της, του εισηγητή, καλωσορίζουμε την προσπάθειά του για να εξασφαλίσει ότι το διοικητικό κόστος ε, να είναι αναλογικό και αιτιολογημένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το πιο ανοιχτό επενδυτικό καθεστώς, να θυμίσουμε. Επίσης, ε, είναι σημαντικό το ότι περιλαμβάνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, δεν θέλουμε επίσης να κάνουμε μαύρες λίστες για κάποιες δικαιοδοσχεσίες, αν και ε, ανησυχούμε για το ότι το Συμβούλιο υποβαθμίζει την αξία αυτή του καταλόγου για φορολογικούς παραδείσους ε, και έχουμε επίσης την ανησυχία ότι πολλές εταιρείε βιτρίνες ε, ε, δημιουργούνται για να διευκολύνουν ευρωπαϊκές εταιρείες να προβούν σε εξαγορές. Πρέπει αυτό λοιπόν να το επανακαθορίσουμε όσον αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις. Όσον αφορά τη δική μας προσέγγιση, λείπουν κάποια στοιχεία από τις προτάσεις της Κομισιόν και του εισηγητή. Το πρώτο είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να απαγορέψουν μια ξένη επένδυση εάν στην χώρα που του προτείνει ισχύει η δικτατορία, δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν συνάδει με τις δικές μας συνθήκες. Επίσης, ε, για τα διάφορα, τους διάφορους ομίλους ή ταμεία θα πρέπει αυτά να τηρούν τις αρχές του Σαντιάγου για τη διαφάνεια και τρίτον δεν υπάρχει ρόλος κανένας εδώ που να προβλέπεται για το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία ελέγχου. Η Κομισιόν θα συλλέγει τις αιτήσεις εκθέσεις των κρατών μελών και θα προβαίνει σε εις βάθος ανάλυση για τις ξένες αυτές επενδύσεις εντός της Ένωσης. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον θα πρέπει να προβλέπετε τακτική έκθεση προς το Κοινοβούλιο για αυτές τις ενέργειες της Κομισιόν, ώστε να και μάλιστα θα πρέπει εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρακολουθεί τις ε, εν λόγω συνεδριάσεις. Ε, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ μόλι και δεν βλέπω άλλους σκιώδεις. Θέλετε κάποιοι να πάρετε λόγο με το ΚΑΤΣΔΙ. Ξέρω ότι η ε, εκπρόσωπος της Επιτροπής από την DigiTrade είναι εδώ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου είμαι τμήματάρχης ε, υπεύθυνη για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, του κυρίου Τσίλε που μας βοηθάει πάρα πολύ. Επειδή ο χρόνος πιέζει θα περιοριστώ σε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, έχουμε την πρόταση για να τροποποιηθεί ο ορισμός του ξένου επενδυτή που θα λέει ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε ξένους επενδυτές ε, επιχειρήσεις ξένης ιδιοκτησίας που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτό είναι αρχή της συνθήκης. Αυτή τη στιγμή μια εταιρεία έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς θεωρείται ευρωπαϊκή. Αν είναι βεβαίως εταιρεία βιτρίνα με μόνο στόχο να παρακάμψει τους ελέγχους, τότε τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο στον κανονισμό μετά υπάρχει μια δεύτερη τροπολογία που αφορά το πώς μπορούν να αποκλειστούν εκ των προτέρων κάποιες χώρες όπως τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Να σας υπενθυμίσουμε εδώ ότι εργαζόμαστε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της αρχής του μάλλον ευνοούμενου κράτους ε, στο, του ΠΟΕ οπότε έχουν υποχρέωση να αντιμετωπίζουμε όλες τις τρίτες χώρες με τον ίδιο τρόπο χωρίς ε, διακριτική μεταχείριση δεν έχουμε εμείς ε, κάποια εξαίρεση ή επιφύλαξη οπότε δεν μπορούμε εκ των προτέρων να εξαιρέσουμε κάποια κράτη αλλά βεβαίως τα κράτη-μέλη όταν κάνουν τον έλεγχο μπορούν να καθορίσουν κριτήρια και αν το να είναι κανείς μέλος του ΝΑΤΟ είναι ένα τέτοιο κριτήριο, οπωσδήποτε μπορεί να ισχύσει για ασφάλεια και δημόσια τάξη, αλλά εκ των προτέρων να αποκλειστούν είναι πρόβλημα όπως είπα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τον λόγο ξανά στον Ρόμπερτ Τσίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημείωσα τις θέσεις σας. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό κάποια πράγματα λίγα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό νομίζω είναι να δούμε αυτό το οποίο είπε η Κομισιόν για κάποια νομικά εμπόδια ε, που δεν τα γνωρίζαμε στον ορισμό αλλά ταυτόχρονα είναι λίγο περίεργο παραδείγματο χάρη ε, στην περίπτωση του πλυντηρίου στον Πάναμα είχαμε επενδύσει από το ένα κράτο στο άλλο και δημιουργούσε την περίπτωση αυτή του πλυντηρίου που λέγαμε των 20 δισεκατομμυρίων. Ε, δεν είναι αυτές άμεσες ξένες επενδύσεις. Ε, νομίζω ότι είμαστε σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Αν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και θα βρούμε κάποιες λύσεις. Αν ε, πραγματικά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ελέγχου το οποίο δεν είναι τόσο καλό σε κάποια μέλη. Σας ευχαριστώ. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα και το πώς θα συνεχίσουμε. Πιστεύω ότι το σχέδιο γνωμοδότηση το συζητήσαμε σήμερα. 7 Φεβρουαρίου, προθεσμία για τροπολογίες, συζήτηση 19 Μαρτίου της τροπολογίας, έτσι ώστε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ 26-27 Μαρτίου και μετά Ολομέλεια. Σε αυτό το χρονοδιάγραμμα ε, πιστεύουμε πως ε, θα περάσει το θέμα. Κλείνει η ζήτηση για το θέμα των άμεσων ξένων επενδύσεων και το επόμενο είναι τα διάφορα. Δεν υπάρχει τίποτα από την Προεδρία και δεν βλέπω κάποιον να ζητάει κάτι. Οπότε κλείνουμε και το σημείο αυτό και το μόνο που χρειάζεται να πω είναι η επόμενη συνάντηση που έχουμε προβλέψει 21 Φεβρουαρίου Τετάρτη 9 με 12.30, 2.30 με 6.30 5.22, 22, 9 με 12.30 Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε θα τα πούμε σύντομα